Euh, Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας εγκρίνοντας την ε, ημερήσια διάταξη. Έχω ένα αίτημα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης από τον κύριο Κάσμαν, ο οποίος θα, ήθελα, θα ήθελε το σημείο 12 να το εξετάσουμε στις 6 Δεκεμβρίου. Μιλούμε για την αναθεώρηση της ε, Συμφωνίας του Κοτονού. Αν συμφωνείτε, δεχόμαστε αυτή την τροποποίηση. Επομένως, ε, καταργείται το σημείο 12 στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη. Θα εξεταστεί στις 6 Δεκεμβρίου. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Λάβατε τα πρακτικά για τις 17 και τις 18 Σεπτεμβρίου του 2012 και αν έχετε παρατηρήσεις επ' αυτών, παρακαλούμε να τα υποβάλλετε στη γραμματεία πριν το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. Ε, οπότε και θα εγκριθούν τα πρακτικά. Τώρα θα υιοθετήσουμε τις αποφάσεις και τις συστάσεις των συντονιστών της 8 η Οκτωβρίου. Λάβατε ε, τις συστάσεις και τις αποφάσεις. Τις έχετε στο φάκελό σας. Εάν έχετε παρατηρήσεις, θα πρέπει να μας τις υποβάλλετε πριν το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. Τώρα, ανακοινώσεις της ε, Προέδρου. Θα ήθελα για τρία λεπτά περίπου να σας μιλήσω για την ε, αποστολή κατά της διαφθοράς, στην οποία και συμμετέχω ως προς το Αφγανιστάν στο πλαίσιο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα πρώτα μου συμπεράσματα. Ε, βεβαίως, θα μεταβώ πάλι στην Καμπούλ από τις 23 Νοεμβρίου μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Η αποστολή αυτή λαμβάνει χώρα με τη συνεργασία δύο διεθνών εμπειρογνωμόνων και τριών Αφγανών εμπειρογνωμόνων εκτός από την υποφαινόμενη για μία περίοδο ε, δύο ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Έχει ως σκοπό να επαληθεύσουμε κατά πόσο υπάρχουν θεσμοί ή θα υπάρξουν θεσμοί που θα μπορούν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στην Καμπούλ. Από τις 7 μέχρι τις 27 Ιουλίου ήμασταν στην Καμπούλ και συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της ε, δημόσιας διοίκησης των επιχειρήσεων, εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και όλοι μας μίλησαν για το πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση ε, του αγώνα της μάχης κατά της διαφθοράς στην ε, Καμπούλ, στο Αφγανιστάν, όπου οι αρχηγοί των φυλών επικρατούν, όπου οι φατρίες επικρατούν και όλα αυτά έχουν προτεραιόνιντα έναντι της δικαιοσύνης. Το Αφγανιστάν έλαβε 28 δις ε, ευρώ ε, βοήθεια από το 2002 μέχρι το 2010. Στη διάσκεψη στο Τόκιο αποφασίστηκε να λάβει 4 δις το χρόνο επιπλέον, άρα 16 δις συνολικά υπό τον όρο ότι θα υπάρξει πραγματικός αγώνας ε, καταπολέμησης της διαφθοράς. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου λάβαμε μια απόφαση η οποία είναι σημαντική κατά τη γνώμη μου να ξεκινήσει μια δημόσια έρευνα για την Καμπούλ ε, Bank η οποία στήχησε εξαιρετικά ακριβά στους ε, Αφγανούς. Η έκθεση αυτή έχει καταρτιστεί, ελπίζω να δημοσιευθεί. Αυτό θα εξαρτηθεί από την απόφαση του οργανισμού μας, ο οποίος ονομάζεται ΜΕΚ. Μπορείτε να βρείτε όλες τις συστάσεις που έχουμε ε, κάνει στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΜΕΚ. Έχουμε καταγράψει και έχουμε καταλήξει σε 57 συστάσεις και το 81% εξ αυτών, ε, για το 81% έχουν υπάρξει αντίστοιχες πράξεις. Π.χ. η εξορρυκτική βιομηχανία οφείλει να δημοσιεύει τις συμβάσεις. Ζήτησε επίσης ένα, ε, να δω ένα στρατόπεδο προσφύγων μαζί με ένα νέο Αφγανό, ο οποίος έφυγε από το Αφγανιστάν όταν ήταν 14 ετών και πράγματι διέσχισε ολόκληρο τον κόσμο. Και θα δείτε στην έκθεση της παρατηρήσεις του. Έχουμε 10.000 εσωτερικούς εκτοπισμένους, εσωτερικού εσωτερικούς πρόσφυγες που ζουν σε κατάσταση απόλυτης ένδυας και ελπίζουμε όλοι βεβαίως ότι η ανθρωπιστική μας βοήθεια θα φτάσει και σε αυτό το στρατόπεδο των προσφύγων. Άλλη ανακοίνωση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξή. Η συνεδρίαση διαπραγμάτευσης για το DCI, ε, το εργαλείο για την αναπτυξιακή συνεργασία, με διακόπτη η γραμματέας, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η συνεδρίαση της Επιτροπής μας την Πέμπτη το απόγευμα ακυρώνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια ανακοίνωση να μας κάνει. Εάν όχι, τότε να πω ότι έχουμε ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκέρενς έχει διατυπώσει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας απαντήσει. Την εκπροσωπεί ο κύριος Άντζελο Μπάγκλιγιου. Πολύ σημαντικά όλα τα ερωτήματα που μας διατυπώνεται, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει γραπτό στο πρώτο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με το θεματικό πρόγραμμα για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση, λέει ο κύριος Γκέρνης. Ως προς ε, το φόρουμ αυτό, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο πολιετές, ενδεικτικό. Δεν θα σας πω τις λεπτομερίες ε, έχουν, υπάρχουν στη γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω όμως να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξής. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει επί τη βάση ποιού έγγραφου ή πάνω σε ποια βάση τύρτισε το πολιετές ενδεικτικό πρόγραμμα και επίσης πώς έλαβε υπόψη της τις τροποποιήσεις που προτείνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για αυτό το θεματικό πρόγραμμα Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό καταρχάς και κατά δεύτερον λόγο μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποια είναι η διαδικασία και πώς φαντάζεται αυτή τη διαδικασία ώστε αυτή η δουλειά της διαβούλευσης και της προετοιμασίας να συμπεριλάβει και τις προόδους που έχουμε επιτύχει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το εργαλείο για την αναπτυξιακή συνεργασία διαπραγματεύσεων που έχουν να κάνουν με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 ε, μια διαπραγμάτευση η οποία βεβαίως συνεχίζεται ακόμα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ωραία. Ο κύριος Γκέρενς μας επανέλαβε τα ερωτήματά του. Κύριε Μπάγκλη, από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εξορισμού ο κύριος Γκέρενς διατυπώνει ε, πολύ ε, έγκριτα και ε, σωστά ερωτήματα. Ως προς το πρώτο ερώτημα θα γνωρίζετε ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου εδώ και δύο χρόνια με το σύνολο ε, των εκπροσώπων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το διάλογο έχει εμπλακεί και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε καταλήξει σε ορισμένες συστάσεις ως προς την τελική δήλωση μετά το σεμινάριο της Βουδαπέστης. Επομένως, επί τη βάση των συστάσεων όλων των εμπλεκόμενων, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε ώστε να καθορίσουμε καλύτερα τις υποθέσεις εργασίας εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Συζητήσαμε πολύ ανοιχτά, όπως το κάνουμε πάντοτε, με όλους τους φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του περασμένου φόρουμ και μάλιστα η κυρία Πρόεδρος μας έκανε την τιμή να παραστεί στην εναρκτήρια συνεδρίαση. Το εγχείρημά μας, η προσέγγιση μας έγκυται στο να κατανοήσουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ανάγκες και πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές με συνένεση μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και πώς ε, μετά από αυτή τη συνένεση θα καταλήξουμε σε προτάσεις δικές μας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, βασιζόμαστε στην ανάλυση των αναγκών, ούτως ώστε να καθορίσουμε μετά τους στόχους της δράσης μας. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει αυτό ε, τη διαδικασία ε, ε, διαθεσμικής, διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Και νομίζω ότι το λέω αρκετά καθαρά στο έγγραφο εργασίας. Είναι προκαταρκτικές προτάσεις αυτές, δεν είναι ακόμα σχέδια συγκεκριμένα. Ε, είναι μια δουλειά που έχει γίνει επί του περιεχομένου. Μόλις οι διαθεσμικές διαπραγματεύσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων ολοκληρωθούν, τότε τα αποτελέσματά τους θα τα λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη ε, προκειμένου να ξεκινήσουμε τη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος. Όποιες και αν ήταν οι επιλογές που έχουν προσδιοριστεί σε αυτή τη διαθεσμική συμφωνία. Είμαστε δηλαδή σε φάση εμβάθυνσης ε, της ανάλυσης για να ε, καθορίσουμε σαφέστατα ποιες είναι οι ανάγκες και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ανταποκριθούμε σε αυτές. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς θέλει να έχει την τελευταία λέξη. Παρακαλώ. Επομένως, αν κατάλαβα καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα νέα στοιχεία που μπορεί τυχόν να προκύψουν μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Έτσι δεν είναι. Ε, έτσι ερμηνεύω την απάντησή σας. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ Α, για άλλη μια φορά και θα ήθελα να εκφράσω τα πιο ε, θερμά συναισθήματα που τρέφω για το πρόσωπό σας. πρώτο σημείο σημαντικό αν θέλετε, στην ε, ημερήσια μας διάταξη είναι πρόταση κανονισμού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ε, σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής ε, Βοήθειας. Είναι μια νομοθετική διαδικασία, εντασσόμαστε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και διαπραγματευθήκαμε με το Συμβούλιο βάσει τακτής διαδικασίας. Ε, το ΕΛΚ έχει καθορίσει, έχει ορίσει την κυρία Μισελ Στρίφλερ ως εισηγήτρια επί της ουσίας και η Επιτροπή για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις θα εκφράσει μια διατυπώση για το θέμα αυτό. Θα ακούσουμε την κυρία Φίνκ Χόγερ, ε, υπεύθυνη επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ, υπεύθυνη για τις στρατηγικές και τις ε, πολιτικές. Θα ήθελα κυρία Χόγερ να σας καλωσορίσω στη δική μας επιτροπή και να σας δώσω ευθύς αμέσως τον λόγο για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για να μας παρουσιάσετε τον πυρήνα της νομοθετικής αυτής πρότασης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ωραία υποδοχή. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να σας παρουσιάσω το πρώτο σημείο της πρότασής μας. Πολύ χαίρομαι που θα τα κάνουμε αυτά μαζί και με την Επιτροπή ΔΕΒΕ που είναι η κύρια Επιτροπή και θα διατυπώσει τη θέση του Κοινοβουλίου στην καινούρια πρόταση. Πολύ καινούρια και μοναδική ευκαιρία είναι αυτή για όλους μας να δουλέψουμε πάνω σε μια πρόταση η οποία ε, προέρχεται από την ε, αλλαγή της συνθήκης και μπορεί να δημιουργήσει μια νέα μορφή έκφρασης αλληλεγγύης της Ευρώπης στα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης χαίρομαι που μπορώ να πω ότι κατά το παρελθόν αυτή η Επιτροπή μας είχε υποστηρίξει και όταν στείλαμε το, την πρώτη ανακοίνωση για να βολιδοσκοπήσουμε προς τα που θα κινηθούμε και ελπίζαμε, ελπίζαμε να μας κάνετε κριτική, αλλά να μας στηρίξετε στην προσπάθεια αυτή. Υπάρχει τώρα μια δυναμική αλλά και χρονικές πιέσεις όπως ξέρετε γιατί η πιλωτική φάση για τους εθελοντές τελειώνει το 2014 και η πολιτική δυναμική του Κοινοβουλίου που βρήκε συμφωνία σε, μια, σε πολιτικό επίπεδο σε μια νέα νομοθετική πρόταση είναι επίσης χρονικά περιορισμένη, δηλαδή πιέζει ο χρόνος. Ελπίζουμε λοιπόν στις αρχές του 2013 να μπορέσουμε να αρχίσουμε συζητήσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου ανάλογα και με το πώς θα πάνε βέβαια οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Εγώ σήμερα θα σας υπενθυμίσω το σκεπτικό, τι έχει υποβληθεί και γιατί. Θα σας δώσω κάποιες ενότητες και θα ακούσω τις ερωτήσεις σας για να απαντήσω. Ε, υποθέτω και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανταλλαγές μεταξύ μας και θα μπορέσουμε να ε, εξειδικεύσουμε την πρότασή μας. Θυμάστε ότι είναι μια πρόταση αυτή που στηρίζεται σε σαφή εντολή από τη συνθήκη της Λισαβόνας Επίσης στηρίζεται σε πολύ προπαρασκευαστική δουλειά, ε, πιλωτική, που την ε, συνεχίζουμε ακόμα και που μας βοήθησε και στις διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο επίσης μαζί σας για να εντοπίσουμε που υπάρχουν ανάγκες και κενά που αυτή η μορφή της νέας βοήθειας με τους θελοντές μπορεί να βελτιωθεί. Πρέπει να βελτιωθεί η ικανότητα της Ένωσης και πρέπει να υποστηριχθεί και η ικανότητα άλλων χωρών ώστε να αντιμετωπίσουν ε, πολλές καταστροφές φυσικές και ανθρωπογενείς. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις δεξιότητες και τα προσόντα των ε, συμμετεχόντων εθελοντών. Αυτή η πρόταση λοιπόν ε, των νέων εθελοντών μπορεί να οδηγήσει σε πιο πολύ επαγγελματισμό στην παροχή της βοήθειας. Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δουλειά αυτή της συνένεσης που έγινε. Βεβαίως στηρίζεται στις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας, βασίζεται στις ανάγκες και στηρίζεται και στο πεδίο εφαρμογής μιας ε, ανθρωπιστικής δράσης. Αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε είναι καλύτερη αποτελεσματικότητα και ποιότητα της βοήθειας μέσα από καλύτερη επιλογή των εθελοντών, πιο καλύτερα εκπαιδευμένων και έτσι θα ενισχυθούν και οι τοπικές οργανώσεις και οι ικανότητες για να έχουμε καλύτερη ε, διατηρησιμότητα, ετοιμότητα στην παροχή της βοήθειας γενικότερα στις τρίτες χώρες. Ήδη ανέφερα τις λέξεις ε, μείωση του κινδύνου καταστροφών, ε, από τελική απόκριση ε, και ανάκτηση της απόκρισης θέλουμε να ε, πληρούνται κενά σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα κυρίως, οπότε σκεφτόμαστε πολύ να τους χρησιμοποιήσουμε στη διαχείριση κινδύνου καταστροφών και στις ε, διαχειριστικές διοικητικές ικανότητες, γιατί υπήρχε εκεί σημαντικό κενό στις υφιστάμενες οργανώσεις. Δεν υπήρχε δηλαδή υποστήριξη back office ε, αν προέκυπταν τέτοιες ανάγκες. Αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν θα σκεφτούμε αναγκαστικά να στείλουμε τους εθελοντές σε πολύ ε, ανασφαλή περιβάλλοντα όταν σκεφτόμαστε για την τιμότητα. Σκεφτόμαστε βέβαια ότι είτε είμαστε σε κατάσταση σε ένα περιβάλλον πριν ή μετά την κρίση. Δημιουργία ικανοτήτων τοπικών κοινωνιών, τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και αυτό είναι ένα θέμα κύριο στην πρόταση γιατί δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε το τοπικό δυναμικό στέλνοντας τους εθελοντές. Αντίθετα, θέλουμε να βοηθήσουμε τους ντόπιου να αναπτύξουν την ε, ικανότητά τους και να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο την εξάρτησή τους από ε, αυτούς και από μας. Κάναμε και μελέτη επιπτώσεων, δεν θα τα πω αυτά όμως γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και επίσης ε, είδαμε και εξετάσαμε κάποιες ε, δυνάμεις που είχαμε στα πλαίσια του πιλωτικού, του pilot. Μέχρι τώρα δύο χρόνια δούλεψε, 214 θελοντές δούλεψαν σε 40 οργανώσεις σε 30 χώρες. Αλλά αυτά είναι πιλωτικά μας δίνουν κάποιες ε, ε, γνώσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι έτσι θα πρέπει να διατυπώσουμε την πρότασή μας, γιατί αν δούμε την ε, πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που υποβάλαμε, είναι ένα σκελετός, ένα πλαίσιο διευκολυντικό αν θέλετε, δεν μπαίνει σε όλες τις λεπτομέρειες. πολλά θα συμπληρωθούν με εκτελεστικές ή κατεξουσιοδότηση πράξη και την επιτροπολογία, αλλά είναι ένα πλαίσιο νομοθετικό, τόσο ώστε να υπάρχει μια βάση για να δομηθούν όλα αυτά, όλε αυτέ οι δομέ. Τέλος, υπενθυμίζω τις διάφορες ενότητες ή θεματικέ. τα δομικά στοιχεία αν θέλετε, για να στηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό για τους εθελοντές. Καταρχήν χρειάζονται πρότυπα πιστοποίηση και ε, πρόγραμμα δημιουργίας ικανοτήτων. Θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ποιοτικό σήμα της Ένωσης, αν θέλετε, για τους εθελοντές, που μετά θα ενσωματωθεί στις υφιστάμενες δομές, στις υφιστάμενες οργανώσεις επιτόπου, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε εκ των προτέρων, πριν αρχίσουμε δηλαδή να τους εκπαιδεύουμε και να τους στέλνουμε, ότι θα έχουμε ικανές οργανώσεις που θα μπορέσουν να αφομοιώσουν και να αξιοποιήσουν τους ε, θελοντές και θα τους ε, στείλουν όπου πρέπει να πάνε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πιστοποίηση. Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν πρότυπα είτε για τη φιλοξενία είτε για την ε, αποστολή και τις οργανώσεις φιλοξενίας και αποστολής. Ε, φροντίδα, η η αξιοποίησή τους, τι είναι σημαντικό σε κάθε τομέα, όλα αυτά ε, που είναι λεπτομέρειες κάθε φορά. Και η δεύτερη ενότητα είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση. Αυτή είναι μία από τις προστιθέμενες αξίες από το πρόγραμμα, ότι θέλουμε να έχουμε εθελοντές που θα είναι αποδοτικοί, έτοιμοι, ε, καλά προετοιμασμένοι, και γι' αυτό θέλουμε να ενθαρρύνουμε συνέργειες μεταξύ υφισταμένων οργανώσεων αλλά και να δημιουργήσουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων και εκπαίδευσης που θα μπορεί να είναι κοινό για όλους. Επίσης μπορεί αυτό να είναι ένα βήμα ενδιάμεσο μεταξύ εκπαίδευσης και ε, πρακτικής δουλειάς για τους νέους ε, και αυτό θα είναι σαν μια μαθητεία μέσα στην Ευρώπη αν θέλετε πριν πάνε να δουλέψουν επί Ίσως όμως πρέπει να πω ότι δεν στοχεύουμε μόνο ε, σε πολύ νέους εθελοντές. Όλες οι ηλικιακέ ομάδες είναι στο στόχο μας, στην ομάδα στόχο και έμπειρους συνταξιούχους θέλουμε, διότι και αυτοί φέρνουν μεγάλη εμπειρία επιτοπίως. Και αν δούμε και τις δημογραφικές αλλαγές, νομίζω ότι θα ήταν ανοησία να μην αξιοποιήσουμε και αυτό το δυναμικό των πιο ηλικιωμένων. Ε, θα έχουμε λοιπόν πρότυπα, θα έχουμε την ε, επιστοποίηση, θα έχουμε ε, την δημιουργία ικανοτήτων και θα δούμε αυτούς που έχουν εκπαιδευτεί, που μπορούν να καταγραφούν σε ένα μητρό για να τους παίρνουν οι οργανώσεις από εκεί και να τους απασχολούν με ένα σύστημα εκπεριτροπής, με βάση ένα εργασιακό πρόγραμμα ε, που θα καθορίζεται από, τους, από τις τοπικές οργανώσεις ή τις οργανώσεις εταίρους μας. Είναι πολύ εταιρικό πρόγραμμα, γιατί ε, η ιδέα δεν είναι να πάρουμε θελοντές από μία οργάνωση ή να κάνουμε διπλή δουλειά, να επαναλάβουμε τη δουλειά που κάνει ο ένας, αλλά να δώσουμε πρόσθετα, προσόντα, πραγματογνωμοσύνη και τοπικά και εδώ. Και στην τελευταία ενότητα κάλυψη αναγκών. Όταν θα έχουμε αυτό το σώμα των νέων εθελοντών για την ε, βοήθεια, αυτοί θα πάνε επί τόπου, θα δουλέψουν εκεί, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσουν πίσω και τότε θα φτιάξουν ένα δίκτυο εθελοντών για να προωθήσουν τον εθελοντισμό, το πρόγραμμα του εθελοντισμού ακόμη περισσότερο. Θα συνεχίσουν επίσης να παρέχουν υποστήριξη ε, και θα έχουμε τη δυνατότητα και online και θα έχουμε δυνατότητα παρακολούθησης. Ξέρω ότι κάποιοι εθελοντές στο τέλος θα μπουν στην αγορά εργασίας και θα είναι και ε, πολύ ε, θα έχει μεγάλη ζήτηση για αυτούς. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Τέλος για τον προϋπολογισμό, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε. Ναι, έχουμε προβλέψει τώρα στο πρόγραμμα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού με 239 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά προφανώς θα εξαρτηθούν από τις συζητήσεις στα πλαίσια του MFF. Ε, έρχεται και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Σύνοδος Κορυφής. Αλλά το αν στο τέλος θα αποσταλούν και θα εργαστούν οι 7 ή 5 χιλιάδες. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε τώρα είναι η 5000 αυτο που πρεπει να δομή, να, αν το νομικό πλαίσιο είναι σωστό, αν είναι σωστό να λύγει και να έχουμε έκφραση αλληλεγγύης και προστιθέμενη αξία, θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με τρόπο ασφαλή και εφικτό και βιώσιμο. Ε, αυτό εννοώ όταν λέω για ένα διευκολυντικό πλαίσιο. Σταματώ εδώ για να απαντήσω και σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην Mrs. Κρίστελ, θέλω να καλωσορίσω το, την ε, ομάδα που μας επισκέπτεται από Γερμανία, από τη Φιλανδία και την Ρουάντα και συμμετέχουν όλοι στην αναπτυξιακή δουλειά. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ για να δείτε πώς λειτουργεί η Επιτροπή Ανάπτυξης. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Να ευχαριστήσω και την κυρία Γεωργίβα, την ε, Επίτροπο, αρμόδια για την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώ και τη Γενική Διευθυνσία, η οποία βοήθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή αυτή τη ε, συζήτηση επί των Ευρωπαίων Εθελοντών Ανθρωπιστική Βοήθειας. Όπω προείπατε, η νομοθετική πρόταση εδράζεται σε ανακοίνωση του 2010. Είχα συμμετάσχει σε κοινή συνέντευξη τύπου με την κυρία Γεωργίευα επί των διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερομένα μέρη και βάση ανάλυση επιπτώσεων. Είχα την ευκαιρία επίσης να συζητήσω κατά επανάληψη με διαφόρους εμπλεκομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ορισμένοι εξέφρασαν του τους δισταγμούς όσον αφορά την ενδεχομένη υπεραξία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και στην σχετική χρηματοδότηση. Ως εισηγήτρια διοργάνωσα με οργανώσεις του τομέα συναντήσεις προβληματισμού επί των προτάσεων της Κομισιόν. Γιατί ότι είναι χρήσιμη η πρόταση. Την Πέμπτη το πρωί θα συναντηθώ με 21 εθελοντές του πιλωτικού προγράμματος υπό τον γαλλικό Ερυθρό Σταυρό. Η ελληνική αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εθελοντισμός είναι έμπρακτη έκφραση, ορατή θα έλεγα έκφραση, αυτής της ελληνικής. Οι Ευρωπαίοι εθελοντές θα αποκτήσουν έτσι εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες, ανεκτήμητες θα έλεγα, που έχει ανάγκη ο πληθυσμό στο πλαίσιο αυτών των αποστολών ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Η πρωτοβουλία συμβάλλει επίση στην ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη και στην προώθηση τη ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Χαίρομαι για το ότι η δράση του σώματος θα διέπεται από τις αρχές μας και ότι η ανάπτυξη του σώματος αυτού θα εξαρτάται από τις συνθήκες. Συγχαίρω την Κομισιόν διότι ο μηχανισμός αυτός συμπληρώνει ήδη φυστάμενες δομές και μηχανισμούς και ότι έχουν αποφευχθεί έτσι οι επικαλύψεις. Καλύπτουμε επίση με τον τρόπο αυτόν και ορισμένα κενά στον τομέα του θελοντισμού. Κατά τη διατύπωση τη εκθεσή μου και των τροπολογιών θα επιμείνω πολύ στα κριτήρια επιλογή των εθελοντών. Η κατάρτιση θα μα επιτρέψει να στέλνουμε κατά τόπου ανθρώπους, ειδικού, επαγγελματίε, για να υπάρχει πραγματικά, όπω είπα, υπεραξία υπέρ των οργανώσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα και εν τέλει υπέρ των ομάδων που έχουν πληγεί από φυσικέ καταστροφέ ή άλλες. Προχωρήσουμε με κατεξουδότηση πράξεις, με γνώμονα επιχειρησιακού στόχου ή με εκτελεστικέ πράξεις όσον αφορά την πιστοποίηση των ε, οργανισμών προέλευσης και προορισμού. Το έτοιμο αυτό τη πρόταση παραμένει αρκετά αόριστο και γενικόλογο όσον αφορά για παράδειγμα την πιστοποίηση των οργανισμών οι οποίοι επιλέγουν του ψηφίου, του καταρτίζουν και εξασφαλίζουν την υποστεμένη αξία. Τι γίνεται ε, για παράδειγμα με την ηλικία κατόφλι των 18 ετών. Αυτά ως προς τις βασικές γραμμές. Κάποιες ε, δράσεις Επίσης θα προκρίνονται μόνο με βάση εκτελεστικές πράξεις. Κύριε Φενκάιλερ, το άρθρο 21 ε, στην παραγραφό 4 ορίζει ότι η Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη της την προσθεμένη αξία και τα πλέον εκτήματα όσον αφορά την διαχείριση που θα προκύψουν από ένα σχετικό ταμείο χρηματοδότησης. Ευχαριστώ για αυτή την διευκρίνηση. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 24, παράγραφος 3, εκεί προβλέπεται η οθέτηση ενό ενιαίου προγράμματος δράσης για την υλοποίηση του κανονισμού. Πώ είναι δυνατόν το πρόγραμμα αυτό, το οποίο προσδιορίζει γενικούς στόχου, ε, γενικά προσδοκόμενα αποτελέσματα και το καθεξής, πώς είναι δυνατόν να ακολουθήσει την επιτροπολογία και όχι τις της πράξης. Σας ευχαριστώ πάντως και πάλι θα συνεχίσουμε την εξαιρετική μας συνεργασία, διότι πιστεύω ότι επί των περισσότερων συμφωνούμε. Θα ήθελα όμω αν είναι εύκολο, να έχω απαντήσεις στα ερωτήματα που μόλις έθεσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Κορτές Θα είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία ξεκίνησε το 2010 με την ανακοίνωσή της, όπως είπε και η κυρία Στρίφλερ. Ως σοσιαλιστές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να πω ότι θα παρακολουθήσουμε εκ του σε αυτή τη διαδικασία. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη διάσταση της ασφάλειας αλλά και της εκπαίδευσης των εθελοντών και επιθυμούμε να εμβαθύνουμε στις ικανότητες και τις αρμοδιότητες αυτών των εθελοντών. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σημαντικό το θέμα, το γνωρίζουμε, αλλά και λεπτό. Κύριε Στρίφερ, έθεσε ευαίσθητα ερωτήματα. Θέλω να τονίσουμε από την πλευρά μου την προσθεμένη αξία της πρότασης. Ξέρετε, για να αποφύγουμε καταρχήν τις επικαλύψεις, Θέλει προσπάθεια. Πριν καν ιδρύσουμε το σώμα, ε, υπήρχαν ανθρωπιστικές παρεμβάσεις. Πρέπει με αυτούς τους ε, οργανισμούς, οργανώσεις, πρωταγωνιστές να έρθουμε σε διάλογο πριν πάρουμε αποφάσεις. Μετά, το θέμα τη ασφάλειας. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ε, ένστολων και μη μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Τι γίνεται λοιπόν όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε ειρηνευτική επιχείρηση. Οι Ευρωπαίοι θελοντές, το νέο αυτό σώμα, θα είναι αρκετά ουδέτερο, αμερόληπτο για να εξασφαλίσει και την ασφάλεια των ακτιβιστών οι οποίοι συμμετέχουν στο σώμα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο περιμένει απάντηση. Και εδώ θα ήθελα η υπηρεσία εξωτερική δράση να μας ενημερώσει, να μας απαντήσει. Διότι τόσο τα κρατημέλη όσο και η υπηρεσία εξωτερική δράσης πρέπει να είναι ουδέτερα. Και θυμηθείτε, δεν είναι μόνο οι φυσικέ καταστροφέ, είναι οι τροπογενείς καταστροφέ, είναι οι πολιτικές καταστροφές, πόλεμοι, όπου μπορεί να απαιτηθεί δική μα δράση και παρέμβαση. Και κάτι άλλο, πάλι για τον σκοπό τη αποφυγή επικαλύψεων. Και συμμερίζουμε αυτό που είπατε εν γέννη, επειδή το θέμα έχει και λεπτομέρειε. Πώ θα χειριστείτε μια έκκληση μιας χώρας η οποία ζητά ανθρωπιστική βοήθεια. Θα δώσετε προτεραιότητα στην χρηματοδότηση και τα συνοδευτικά μέτρα σε αυτούς που συμμετέχουν στο σώμα, που έχουν δηλαδή πιστοποίηση, αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της πιστοποίησης, και εμπροκειμένο και κατά συνέπεια μόνο σε δεύτερο χρόνο θα μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων που δεν έχουν πιστοποίηση. Το λέω αυτό για να μην προκύψουν αντιπαραθέσεις μεταξύ των ίδιων οργανωμένων ανθρωπιστικών οργανώσεων που, υπά, που υφίστανται αυτή τη στιγμή και των άλλων. Οπότε, επαναλαμβάνω, πώς θα δημιουργηθεί και πώς θα λειτουργήσει αυτό το σώμα. Κυρία Στρίφερ είπε στην εισαγωγή της και εγώ θα πω με τα δικά μου λόγια τι θέλετε να αποφασιστεί στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Μπορεί να φαίνεται η ερώτηση, αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να το διευκρινίσουμε αυτό τώρα μέσως. Τι, θα, τι από την συνεπόφαση. Εάν φύγουν οι στρατηγικές προτεραιότητες. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει του 290 και του 291, δεν θα διαδραματίσει το ρόλο που του αρμόζει. Ευχαριστώ. Ρος, στην Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας, γιατί είναι ενθαρρυντικό να ακούμε συγκεκριμένες και επικοδομητικές ερωτήσεις, γιατί μας βοηθούν και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. στο οποίο κάναμε μια παρουσίαση και ε, συζητούμε τώρα τα περισσότερα άρθρα. Λοιπόν, οι πολύ σόφρονες ερωτήσεις ε, της κυρίας Στρίφλερ για το διευκολυντικό πλαίσιο. Πολλά θέματα και δράσεις θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τους εθελοντές. Αυτό θα προσδιοριστεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που θα στηριχθεί στην Επιτροπολογία. Δώσαμε παραδείγματα μέχρι τώρα όπως διαχείριση κινδύνου, καταστροφών, διοικητικές, διευθυντικές ικανότητες και η δημιουργία τους και τα συναφή. Αυτά είναι ενδεικτικά και με βάση την εμπειρία που είχαμε από το πιλωτικό. Όμως έχουμε και ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και εντάσσονται αυτά εκεί. Το πρώτο μέλημα είναι να υπάρξει σωστή βάση και λειτουργικό πλαίσιο, γιατί Ποιο ξέρει τι δράσεις θα χρειάζεται δύο ή τρία χρόνια. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές μακροπρόθεσμα στις καταστάσει. και γι' αυτό ένα πρόγραμμα εργασία είναι καλύτερη πρόταση. Προφανώς μπορούμε να δώσουμε και παραδείγματα, αλλά ίσως δεν πρέπει να είναι εξαντλητικά τα παραδείγματα αυτά στην νομοθετική πρόταση. Έχουμε απαριθμίσει παραδείγματα στο προήμιο, όπως λέγεται, όπου δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ε, δημιουργία αντοχής, ε, ετοιμότητα πρόληψη, όχι τόσο στην αντίδραση. Υποδηλώνει κάποια πράγματα, δίνει κάποιες ενδείξεις, αλλά ε, όχι πολλά σε αυτά τα πλαίσια. Εμείς θα εξειδικεύσουμε τις δράσεις σε αιτήσια βάση μέσα από το πρόγραμμα εργασίας. Και έτσι θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε ανάλογα και την εκπαίδευση. Βέβαια, χρειάζεται κάποια βάση ε, ή ένα πακέτο εκπαίδευσης κατάρτισης, το οποίο χρειάζεται όπου και να πάει να δουλέψει κανείς. Μια βασική εκπαίδευση που θα καλύπτει τις αρχές ε, της ομοφωνίας, τις πρώτες βοήθειες, τέτοια πράγματα πολύ βασικά. Ε, ακούγονται ίσως κοινότοπα που πάντως θα πρέπει να υπάρχουν. Και μετά θα εξατομικεύσουμε τις ανάγκες και την εκπαίδευση στις ανάγκες ανάλογα με το που θα πάνε να δουλέψουν και για να αντιμετωπίσουν και τα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευόμενου. Γιατί όπως είπα δεν στοχεύουμε μόνο στους νέους ανθρώπους που είναι και, θα είναι και άπειροι, αλλά και στους έμπειρους που μπορεί να έχουν εμπειρία από το πώς θα τρέξει ένα πρόγραμμα υποδομών ή ένας καταβλισμός που θα μπορούσαν να να μας βοηθήσουν να βοηθήσουμε μια τρίτη, χώρα να προετοιμαστεί καλύτερα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ε, τώρα, για τα καταπιστεύματα. Και αυτό είναι μια διευκολυντική ρήτρα που έχουμε συμπεριλάβει. Γιατί όπως ξέρετε, στο, και στον τωρινό και στο μελλοντικό δημοσιονομικό κανονισμό θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοια ε, ταμεία καταπιστεύματα για την ανόρθωση κάποια χώρα. Αυτό για χώρες που δεν έχουν μεγάλο προϋπολογισμό μέχρι τώρα στην ανθρωπιστική βοήθεια, που μέχρι τώρα συμμετείχαν λιγότερο, αλλά που θέλουν να διοχετεύσουν πόρους και να συμβάλλουν στην παροχή της, Ευρωπαϊ... της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να διοχετεύσουν κάποια κονδύλια μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας των εθελοντών μέσα από την Κομισιόν. Αυτό συνδέεται πολύ από το πώς θα ερμηνεύσουμε και θα συστήσουμε αυτή τη νέα δυνατότητα στα πλαίσια του καταπιστεύματος. Δεν θέλουμε όμως να αποκλείσουμε αυτή τη δυνατότητα από την πρότασή μας, γιατί ανοίγει καινούργιες ευκαιρίες. Και όλοι ξέρουμε ότι θα έχουμε λιγότερα χρήματα στο μέλλον, και άρα θα πρέπει να κάνουμε με τα λιγότερα περισσότερα. Και μπορεί αυτά τα ειδικά ταμεία όρθωση των χωρών, ε, τα καταπιστεύματα, να βοηθήσουν. Γι' αυτό θα τα ε, εντάξουμε. Πολύ σωστά μιλήσε, αναφερθήκατε στην ασφάλεια. Αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ στις συζητήσεις με τους εμπλεκομένους. Γιατί προφανώς δεν ε, ε, θέλουμε αυτούς τους νέους εθελο, τους, ε, το σώμα των εθελοντών και αυτό είναι και μια ανησυχία του κυρίου Γκέρενς νομίζω. Δεν θέλουμε να τους κάνουμε ένστολους και να τους στέλνουμε σε καταστάσεις ε, απρόβλεπτες και, κατε, και κατεπίγουσες και μάλιστα δεν λέγεται πια σώμα. Δεν θα εκφράζουμε αυτή την ιδέα δηλαδή ότι δημιουργούμε ένα σώμα που θυμίζει στρατό. Όχι. Είναι η εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολίτες που θέλουν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους συμμετέχοντας σε κάτι το οποίο ε, είναι πολύ ψηλά στην προτεραιότητα των ευρωπαϊκών αξιών. Και υπάρχει ήδη. Δεν είναι δηλαδή ένα σώμα ανεξάρτητο, αυτόνομο. Οπότε και από την άποψη της ασφάλειας, όποτε τους στέλνουμε και η και η οργάνωση της αποστολής και η οργάνωση της φιλοξενίας θα πρέπει να, πληρεί, να ε, πολλές παραμέτρους ασφαλείας. Και αυτό ακούγεται κοινότοπο, όπως ας πούμε να έχουν ένα πρόγραμμα ασφάλισης, η κάλυψη να έχουν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά να μπορούν και να τους ε, στέλνουν πίσω. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να παρακολουθούμε από κοντά την απασχόλησή τους εκεί και να δούμε πού πρόκειται να εργαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Η ασφάλεια όμως είναι πολύ ψηλά στην, ε, στις προτεραιότητές μας και όταν θα ζητήσουμε προτάσεις και όταν θα μιλήσουμε για την πιστοποίηση των οργανώσεων φιλοξενίας και αποστολής. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που συνδέονται και με την προστιθέμενη αξία και το που θα εργαστούν, που θα απασχοληθούν σε ένα περιβάλλον ασφαλείας. Ε, η αντίδραση είναι μια δυνατότητα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το προ και μετά της καταστροφής, είτε αυτή είναι φυσική είτε ανθρωπογενής. Μας ενδιαφέρει το πριν και το μετά. Δεν αποκλείουμε όμως, και γι' αυτό έχουμε αυτή τη διευκολυντική ρήτρα, δεν αποκλείουμε, εάν χρειαστεί κάποια ικανότητα, για τα ίδια τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της ΕΚΟ, σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν εθελοντές πολύ καλά καταρτισμένη. Πάλι μια διευκολυντική ρήτρα θα είναι αυτή, την οποία πρέπει να δούμε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας. Η πρόληψη και η ετοιμότητα και η διαχείριση του κινδύνου του, της καταστροφής είναι και εν πολλής ανθρωπιστική δράση. Κάποιοι μπορεί να πούν να είναι διαχείριση κινδύνου καταστροφών. Άλλοι μπορούν να πούν σύνδεση της αποκατάστασης με την ανακούφιση, τη βοήθεια. Ε, πάντως, ε, το βασικό σε όλα αυτά είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ε, παρεμβάσει και με βάση την ετοιμότητα. Επίσης, πολλές φορές οι τοπικές κοινότητες δεν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένε και ετοιμασμένες. Ε, επίσης, ε, μια ερώτηση, ας πούμε, εάν συμβεί κάτι σε μια κατεπίγουσα ανάγκη, Πού θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση. Πολύ θεμητό το ερώτημα. Και γι' αυτό ετοιμάσαμε χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού. Διότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για τη σύσταση αυτών των εθελοντών, της ομάδας των εθελοντών, και βέβαια στην αρχική φάση προφανώ θα έχουμε υψηλότερε δαπάνε. Όταν στηθεί το πρόγραμμα και τρέχει θα είναι πιο εύκολο να προβλέπουμε τι δαπάνε. Αλλά το αρχικό κόστο για το, τον οργανισμό, για να δημιουργηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευση, για να υπάρξουν τα πρότυπα, να καθοριστούν κλπ. Αυτό θα απαιτήσει πιο πολλά χρήματα στην αρχική φάση. Και μετά θα πάνε να δουλέψουν εκεί. Γι' αυτό όμω προβλέπεται χωριστή γραμμή του προπολογισμού. Γιατί αν υπάρξει κάτι κατεπήγον, δεν θα μπορέσουμε να, λειτου... να πάρουμε ε, δάνεια, η επιχειρηματικά δάνεια αν θέλετε, για να μειώσουμε την ικανότητα ε, απόκρισης ε, με ανθρωπιστική βοήθεια σε μια κατεπίγουσα κατάσταση και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα δώσουμε αυτά στους εθελοντές. Όμως ε, Αυτό είναι το καθημερινό ψωμί της δουλειάς του ΕΚΟ. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους εταίρους μας, τους ε, FPA εταίρους μας, που θα είναι πιστοποιημένοι, όχι όλοι, κάποιοι όμως θα είναι, ούτως ώστε να μπορούν να δράσουν ως ε, οργανώσεις αποστολής. Για την επιτροπολογία νομίζω ότι θα χρειαστεί μια πιο μακρά συνεδρία. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν καλά. Ε, α, για την ορατότητα και τις στολές έγινε μια ερώτηση. Δεν είναι αυτό το βασικό μας, όπως σας είπα. Δεν θα, τα τους στείλουμε στο Αφγανιστάν ή τώρα στη Συρία. Θα τους στείλουμε ίσως τους ε, ε, καταβλισμούς των προσφύγων στις γειτονικές χώρες, όπου χρειάζονται κάποιες διευθυντικές ικανότητες για να λειτουργήσει ένας καταβλισμός. Κάτι τέτοιο θεωρητικά θα μπορούσα να φανταστώ ε, για τους εθελοντές. Εκεί θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τις υφιστάμενες οργανώσεις που είναι λίγο ε, αδύναμες σε ό,τι αφορά τις διαχειριστικές τους ικανότητες, αλλά δεν θα τους στείλουμε στη, πρώτη γραμμή του πυρός και η ορατότητα που θέλουμε να τους δώσουμε ε, δεν ε, είναι κάτι ιδιαίτερο στις προτεραιότητές μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκιόρενς και μετά η κυρία Στρίφλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως προς την Επιτροπολογία, θα ήθελα να διευκρινίσω στους επισκέπτες μας από τη Ρινανία Παλατινάτο ότι επιτροπολογία σημαίνει ε, ο, χώρος όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πλέον καθόλου λόγο. Ε, στις κατεξουσιδότητες πράξεις έχουν ε, ίδιο βάρος το λόγο τους και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ναι, λοιπόν. Η απάντηση ήταν αρκετά ε, ασαφής και γι' αυτό εκφράζω την απογοήτευσή μου. Το ερώτημα δεν το απευθύνουμε μόνο σε εσάς απευθύνεται και στο Συμβούλιο κατά κύριο λόγο, το οποίο οφείλει να συμφωνήσει μαζί μας για το πώς θα μοιραστούν οι ευθύνε. Και θα ήθελα να ακούσω από πλευρά Συμβουλίου ε, μία πρώτη απάντηση, έστω προσπάθειας απα, απάντησης για το ε, για ποια θέματα θέλουν να υπάρχει ε, ίσο βάρος, αν θέλετε, ίδιο βάρος στο λόγο μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ας προσπαθήσει ε, να το απαντήσει το ερώτημα αυτό το Συμβούλιο και αν πρέπει να καταβάλει τεράστια προσπάθεια, προσπαθήσει να υποβάλει και γραπτή απάντηση. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, εκπροσωπείται το Συμβούλιο εδώ στην Επιτροπή μας. Υπάρχει εκπρόσωπος. Ε, εσείς, παρακαλώ. Πράγματι, και εγώ δεν καλύφθηκα ως προς το ερώτημα περί επιτροπολογίας και συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Γκέρενς. Θα πρέπει να έχουμε κάτι πολύ πιο στέρεο στα χέρια μας πριν δουλέψω πάνω σε αυτή την έκθεση. Ως προς τους εθελοντές, εγώ δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να αποστέλουμε εθελοντές σε ζώνες σύγκρουσης. Νομίζω ότι ήδη είναι αρκετές οι φυσικές καταστροφές, τα στρατόπεδα, οι καταβλισμοί προσφύγων τις περιοχές αυτές, ώστε να μην χρειάζεται να στείλουμε και άλλους ανθρώπους εκεί, εθελοντές μάλιστα. Έτσι βλέπω τα πράγματα, δεν βλέπω πώς άλλος μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Φινκ Χόγερ, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη έχω πει, ωστόσο χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις ε, ως προς την επιτροπολογία από την πλευρά σας. Είναι κάτι στο οποίο επιμένουμε ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Ένα λεπτό μόνο, γιατί έχουμε λίγο καθυστερήσει, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε προβλέψει στην πρόταση, στο άρθρο 9, το οποίο έχει να κάνει με τα πρότυπα και μάλιστα ασφάλειας μεταξύ άλλων, ότι θα δουλέψουμε εκεί με εξουσιοδότηση πράξης. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της θα δουλεύει. Ενώ στο άρθρο 10 έχουμε επιστοποίηση, μηχανισμός, ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, ε, πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εκεί θα δουλέψουμε με εφαρμοστικές πράξεις στο άρθρο 10. Αυτή είναι η πρότασή μας. Μόλις τώρα ξεκίνησε η συζήτηση με το Συμβούλιο. Για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να πούμε ότι το Συμβούλιο δεν έχει καν υιοθετήσει καμία θέση, θέση για το θέμα αυτό. Αλλά τους ενδιαφέρει το ζήτημα και εμείς είμαστε ανοιχτοί ε, προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλουμε να ακούσουμε τους πάντες. Είναι πολύ νωρίς στη διαδικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη δική μας πρόταση τα θέματα αυτά καλύπτονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 10. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, για αυτή την πολύ διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας μας διάταξης ε, συμφωνία Αλλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ζεζίν Μάισνερ. Πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή μας είναι κατά της, της συμφωνίας αλλιευτικής σύμπραξης με τη χώρα αυτή εδώ και δύο χρόνια λόγω των γεγονότων που έχουν σημειωθεί ε, στη χώρα αυτή, τη Γουινέα Μπισάου. Θα δώσω το λόγο όμως στην κυρία Μάισνερ για να μας παρουσιάσει την άποψή της. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι η Γουινέα Μπισάου τώρα δεν έχει νόμιμη κυβέρνηση. Τον Απρίλιο του 2012 έγινε πραξικόπημα στρατιωτικό. Από τότε υπάρχει μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο και μεταβατική κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ούτε διεθνώς ούτε από την Ένωση. Και υπήρξε και ψήφισμα του Κοινοβουλίου που καταδίκασε το στρατιωτικό πραξικόπημα, όπως και τα Ηνωμένα Έθνη που κάλεσαν τη Γουινέα Μπισάου να κάνει δημοκρατικές εκλογές και να ξαναγυρίσει την ομαλότητα. Τώρα όλες οι σχέσεις ε, Ένωση Ουινέα Μπισάου ε, βρίσκονται σε αναστολή, έχουν διακοπή. Έτσι λοιπόν δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Γιατί αν πούμε θέλουμε δημοκρατική κυβέρνηση και δημοκρατική κυβέρνηση δεν υπάρχει, τι να κάνουμε. Ε, μπορεί, αν θα υπάρξει νέα δημοκρατική κυβέρνηση, θα χρειαστούν νέες διαπραγματεύσεις και να εκπέσει αυτή η πρόταση. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Αλληλείας. Θα το σκεφτούν λοιπόν, θα το συζητήσουν και πολύ πιθανό είναι να αναβάλουν την ε, συμφωνία. Βέβαια δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ε, θα πούμε ότι λύγει το θέμα ή θα ασχοληθούμε με αυτό. Αυτά ήθελα να σας πω εξ αρχής. Τώρα, για τη συμφωνία καθ' αυτή, η Γουινέα Μπισάου είναι από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και εξαρτάται από τη βοήθεια πάνω από το 80% του κρατικού προϋπολογισμού είναι υποστήριξη από το εξωτερικό. Στο δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών είναι στη θέση 176 από συνολικά 187 χώρες και αυτό τα λέει όλα. Και πράγματι η αλληλεία για τη Γουινέα Μπισάου είναι πολύ σημαντική. Έχουν και γεωργία, κάσιους ε, ε, ξηρούς καρπούς παράγουν, αλλά η, τα ψάρια είναι η βασική του στροφή. Και τώρα, όπως σας είπα, λόγω της μεταβατικής κυβέρνησης και της τωρινής κατάστασης, βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση εκεί. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλει να αλλιεύει στη Γουινέα Μπισάου που έχει τόσο πλούσια αποθέματα αλλίας και γι' αυτό θέλει και υπήρχε και κατά το παρελθόν η συμφωνία που 17 Τρίτου του 2008 τέθηκε σε ισχύ με τη χώρα αυτή και διάφορα πρωτόκολλα και ε, τώρα είχε αναλάβει η Κομισιόν το, την εντολή να ε, διαπραγματευτεί καινούρια ε, συμφωνία, γιατί η προηγούμενη έληξε. Και τώρα όμως είμαστε σε αυτή την κατάσταση λόγω της ε, ε, ιδιαιτερότητα ε, της πολιτικής. Επίσης η αλία είναι πολύ σημαντική για την Γουινέα Μπισάου. Γενικά μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι έχει νόημα όταν ε, με το καλό θα επανέλθει η ομαλότητα και η δημοκρατική κυβέρνηση να συναυθεί μια νέα συμφωνία και γενικά μπορούμε να συμφωνήσουμε ή να απορρίψουμε. Εν πάση περιπτώσει η εντολή θα πρέπει να δοθεί. Εγώ διαπίστωσα στη γνωμοδότησή μου ότι δυστυχώς υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μου αρέσουν και τόσο πολύ από άποψη αναπτυξιακής πολιτικής όπως ήταν στην προηγούμενη συμφωνία. Δεν ζητάνε διαφάνεια για παράδειγμα στα κονδύλια πώς θα δαπανώνται αυτά που τους δίνουμε εμείς, δηλαδή πώς θα τα δαπανούν. Στην προηγούμενη συμφωνία ήταν καλύτερα ρυθμισμένα αυτά τα θέματα. Υπήρχε και ένα άρθρο 12 στην προηγούμενη συμφωνία που έλεγε ότι το πρωτόκολλο μπορεί να ανασταλεί αν δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις τους, αν για παράδειγμα η βιώσιμη αλληλεία, η αηφόρος δεν ε, τηρείται και η βιώσιμη αλληλεία είναι βέβαια θέμα της Επιτροπής αυτή την απασχολεί. Αλλά και από αναπτυξιακής πολιτικής μπορούμε να σκεφτούμε πόσο σημαντική είναι η αλληλεία για τη χώρα αυτή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει και μια πτυχή αναπτυξιακής πολιτικής. Επίσης θα πρέπει να πούμε στην συμφωνία αυτή την οποία είπαμε κάποια στιγμή αργότερα. Κατά πάσα πιθανότητα θα διαπραγματευτούμε να πούμε ότι είναι σημαντικό το ανώτατο όριο ε, του επιτρεπτού για βιώσιμη αλία να μην υπερβαίνεται μέγιστη διαρκή απόδοση και να ε, ρυθμιστούν τα θέματα των ποσοστώσεων για την ε, ε, ντόπια αλληλεία. Υπάρχουν πράγματα που είναι καλά. Οι περισσότεροι που ε, ψαρεύουν εκεί στους πλούσιους ψαρότοπους δεν είναι ντόπιοι, αλλά υπάρχουν όλο και περισσότεροι ντόπιοι που εργάζονται στα κοινοτικά σκάφη και έχουν καλές συνθήκες εργασίας δηλαδή εκεί. Αυτά έχω να σας πω προς Είναι σημαντικό να γίνει συμφωνία. Αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί οι σχέσει, και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε. Αλλά πάντω ήρθε η ώρα εμεί να γνωμοδοτήσουμε σήμερα και υπ' αυτή την έννοια πήρα και εγώ θέση να υπογράψουμε μεν, αλλά να εκφράσουμε και ορισμένε επιθυμίε και αιτήματα σε σχέση με το τι είναι σημαντικό για την Κομισιόν για να ευημερούν και οι άνθρωποι εκεί επιτόπου. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεβίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Μάισνερ για την πολύ καλή σας έκθεση. Πολύ σημαντικά πράγματα να στην έκθεσή σας. Ιδιαίτερα η υποβάθμιση αυτής της συμφωνίας σε σχέση με την προηγούμενη που με εκπλήσει και λιγάκι γιατί υποθέταμε ότι έπρεπε να γίνει το αντίθετο, να είναι καλύτερη συμφωνία η τωρινή. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από την Κομισιόν εδώ, δεν βλέπω. Πώς γίνεται Θέλω να του ρωτήσω, πώς γίνεται δηλαδή να, για την κατανομή οικονομική βοήθεια, τομεακή βοήθεια, να έχουν λιγότερε υποχρεώσει εκεί στη Γουινέα Μπισάου και λιγότερε υποχρεώσει ό,τι αφορά την ανάπτυξη του τομέα τη Αλία. Τώρα, για την σύναψη συμφωνία πριν εκλεγεί δημοκρατική κυβέρνηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα έπρεπε να συμφωνήσει πριν να έχουμε κάποιο συνομιλητή από εκεί νόμιμο, νομιμοποιημένο, αυτό είναι παράλογο. Και θα, αν γινόταν θα έστελνε εντελώ λάθος μηνύματα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στη Γουινέα Μπισάου. Δηλαδή, τι μήνυμα θα αποστείλουμε, ότι εμείς θα κάνουμε συμφωνίες με όποιον λάχη να ε, ε, κρατάει τα ε, νία της κυβέρνησης, μη νόμιμα. Αύριο το πρωί θα γίνει συνάντηση των συντονιστών στην Επιτροπή Αλίας και αυτό το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξή τους. Ελπίζω, χωρίς να είμαι βέβαιη, ελπίζω όμως ότι θα ε, συμφωνήσουν να αναβληθεί η όλη εξέταση της συμφωνίας. Δυστυχώς, ε, ο θέλει να γίνει και να είμαστε έτοιμοι όταν θα υπάρξει νέα κυβέρνηση, αλλά είναι παράδοξη λογική, γιατί συνήθως δίδουμε συγκατάθεση σε αυτές τις συμφωνίες αφού έχουν συναυθεί και έχουν υλοποιηθεί. Και μάλιστα αυτό πολλές φορές το επικρίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι μας έρχεται συμφωνία αφού ε, έχει ήδη ε, τεθεί σε ισχύ μετά από 8-9 μήνες. Θυμάστε με το Μαρόκο τι έγινε. Ήταν ένα παράδειγμα, ότι πήραμε τη συμφωνία και δώσαμε συγκατάθεση εκ των υστέρων ενώ εδώ θα είναι πρωτοφανές το περιστατικό στη συμφωνία όπου καλούμεθα να συμφωνήσουμε σε μια συμφωνία αλληλείας <clears throat> πριν να συναυθεί. Άλλωστε και το Συμβούλιο ε, σταμάτησε να ε, επεξεργάζεται τη συμφωνία. Θα ήταν εντελώς λάθος μήνυμα από το Κοινοβούλιο κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή Ανάπτυξης θα μπορούσε απλώς να αρνηθεί, να γνωμοδοτήσει πώς θα το χειριστούμε. Και επίσης και η Επιτροπή Προϋπολογισμών με κάνει να αναρωτιέμαι, γιατί και αυτοί συνήθως γνωμοδοτούν επί όλων των αλλιευτικών συμφωνιών. Δεν ξέρω, κυρία Μάισνερ, τι ξέρετε για αυτό το θέμα, τι κάνουν εκείνοι εκεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Λοιπόν, έτσι το βλέπω εγώ το θέμα. Τώρα, επί της ουσίας, μια σύντομη παρατήρηση Μιλήσατε για την εμπορία ναρκωτικών, στο το εμπόριο ναρκωτικών που η Γουινέα Μπισάου πάει να γίνει κέντρο μεταφόρτωσης από την ε, Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Για μένα και γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η αλληλεία για τον προϋπολογισμό της Γουινέας Μπισάου, είναι 7,8% του κρατικού προϋπολογισμού και εσείς είπατε 88% του προϋπολογισμού της, ε, των δαπανών ε, για τη συναλλία προέρχεται από τις συμφωνίες Αλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε αυτά τα πλαίσια αυτό που κάναμε όταν ε, δώσαμε συγκατάθεση για το προσωρινό πρωτόκολλο, το μεταβατικό, αυτό που θα άρχιζε τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, και έπρεπε να σταματήσει λόγω του πραξικοπήματος, νομίζω ότι ήταν δικαιολογημένο με την έννοια ότι θέλαμε να στηρίξουμε μια σταθερή κυβέρνηση και να αναγνωρίσουμε και ότι είναι πολύ μεγάλη πηγή εισοδήματο η αλληλεία στη Γουινέα Μπισάου. Αλλά η Συμφωνία Αλληλεία πρέπει να εφαρμοστεί σωστά ει ό,τι αφορά την αηφορία, την περιβαλλοντική, τα δημοκρατικά δικαιώματα. Και εδώ πόρο απέχουμε από το σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ε, ερωτώ λοιπόν, μπορούμε να αρνηθούμε να γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή Ανάπτυξης πώς γίνεται, τι, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Στρίφλερ. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι η δήμον επί της Αλίας. Εξ όσων γνωρίζω νομίζω, έχω την αίσθηση, γιατί το συζητήσαμε και με τον κύριο Πόγκια, τον ειδικό για την Αλία, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο όλο αυτό τον καιρό η βιώσιμη αλία, η υπεύθυνη αλία και θεωρώ ότι αυτές οι συμφωνίες σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν με τις δικές μας επιθυμίες στην Επιτροπή για την Ανάπτυξη. Εγώ συμφωνώ λοιπόν με τους Πρασίνους και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Να μεταθέσουμε τη θέση σε ισχύ αυτής της συμφωνίας δεν είναι κάτι που επήγει. Εάν με αυτή τη συμφωνία έχουμε ακόμα λιγότερες εγγυήσεις από αυτές που είχαμε πριν, τότε τι νόημα έχει αυτό οι μικρές χώρες ε, δεν θα μπορούν ποτέ να βγουν από αυτήν. Δεν θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας από τη μία και από την άλλη να επιβάλλουμε όλο και λιγότερο αυστερούς κανόνες. Βέβαια, οι συντονιστές δεν είναι εδώ, αλλά εγώ είμαι υπέρ της ε, πρότασης των πρασίνων. Δεν ξέρω, ο Μωρίς τι πιστεύει. Κύριε Πόγκα, έχετε το λόγο. Πόγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ προς την ίδια κατεύθυνση κινούμε ως προς τη Γουινέα Μπισάου, η οποία δεν έχει καθόλου σταθερή και αιρετή κυβέρνηση. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου σταθεροποιηθεί αυτή η χώρα και διενεργηθούν ελεύθερες εκλογές με διαφάνεια και στη συνέχεια βεβαίως να τεθεί σε ισχύ αμέσως συμφωνία αλλιευτικής σύμπραξης. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο. θα πάρω και εγώ το λόγο ένα λεπτό για να πω ότι και στην Αλία, όπως και για όλους τους άλλου τομεί του οποίου εξετάσαμε με τον κύριο Σβένσον, δηλαδή το εμπόριο για την ανάπτυξη, ε, βασικό μας μέλημα δεν θα πρέπει να είναι μόνο η πρόσβαση της Ευρωπαϊκή Ένωσης στους πόρους, στις πρώτες ύλε. Βεβαίως ε, μας ε, πιέζουν να δράσουμε γρήγορα για να αποκτήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Αλλά εμείς κινούμαστε και με άλλο γνώμονα και δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή τη συμφωνία έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή. Καλώς. Να δώσω τώρα το λόγο την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ισαμπέλ Βιαλόν ή στην εκπρόσωπο κυρία Μαρία Μολίνη. Εσείς διαλέγετε, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι παρόντα εδώ. Πρώτον, να σας μιλήσω για το πολιτικό πλαίσιο και δεύτερον, για την έκθεση αυτή καθεαυτή. Τώρα, ως προς την πολιτική κατάσταση στη Γουινέα Μπισάο, τον περασμένο χειμώνα κάναμε τη διαπραγμάτευση για το πρωτόκολλο και τη μονογράψαμε πριν από το πραξικόπημα. Βεβαίως μετά έγινε πραξικόπημα και άλλαξε ε, άρδινη κατάσταση. Όπως ε, το, μας το είπε και η κυρία Λεβίν, το Συμβούλιο εξέτασε από τεχνική σκοπιά στο έγγραφο, αλλά ανέστηλε την ε, λήψη απόφασης λόγω της πολιτικής κατάστασης στη χώρα αυτή. Δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις για την προσωρινή εφαρμογή τέτοιου πρωτοκόλλου. Δεν είχαμε λοιπόν επίσημη, ε, επίσημο διάβημα προς το Κοινοβούλιο από πλευρά Συμβουλίου. Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από τα, τις τελευταίες ε, εξελίξεις που ε, μας είπε η αποστολή που έχουμε επιτόπου είναι το εξής. Όσο περισσότερος χρόνος κυλάει, τόσο λιγότερο είναι οι πιθανότητες να τεθεί σε ισχύ αυτό το πρωτόκολλο. Αυτά από πλευράς πολιτικού σκηνικού. Τώρα, επί της ουσίας, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια σύγχυση ή ασφαλμένη ερμηνεία. Ε, θέλω να επιμείνω στο εξή. Αντιθέτως, το πρωτοκόλλο αυτό με το άρθρο 3 και το άρθρο 12 αυτό που κάνει είναι να ενισχύει την αιρεσιμότητα, της ε, βοήθειας που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στο άρθρο 12 απαριθμούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες εάν δεν πληρούνται ε, υπάρχει κάθε δυνατότητα να ανασταλεί η βοήθεια που δίνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις ή δεν εκτελούνται τα συμπεφώνηθέντα. Και αυτός ήταν ένας και από τους στόχους της μεταρρύθμισης της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής έχουμε προβλέψει ένα νομικό ε, μέσο ούτως ώστε να μπορούμε να αναστέλουμε τις πληρωμές σε περίπτωση μη εκτέλεσης των συμπεφωνδιθέντων. Έχουμε δηλαδή δυνατότητες ε, στη διάθεσή μας ικανοποιητικές. Θέλω λοιπόν να καθησυχάσω τα μέλη της Επιτροπής και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη τεχνική λεπτομέρεια. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, η κυρία Μάισνερ θα πει την τελευταία λέξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, ε, έχω κάπως διαφορετική ανάγνωση. Ήθελα κάτι διαφορετικό σε διατύπωση ε, για το για την ουσία βεβαίως μας ενδιαφέρει από αναπτυξιακή ε, πλευρά και για τη διαδικασία είπα ότι είναι πολύ παράδοξη και τρελή κατάσταση να γνωμοδοτώ σήμερα σε, επί μιας συμφωνίας που δεν μπορεί να συναφεί. Καν θεωρώ εγώ γιατί δεν έχει νόημα. Αφού δεν υπάρχει αναγνωρισμένη κυβέρνηση, πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι θα συνάψουμε μαζί τους συμφωνίες. Αυτή όμως είναι η κατάσταση. Τώρα ε, έχει προγραμματιστεί, σήμερα έπρεπε να το δούμε. Δεν ξέρει και η κυρία Λουβίν τι θα γίνει αύριο. Εγώ ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι να προτείνω αναβολή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως προϋπόθεση θέτει την τη διαπραγμάτευση με τις δημοκρατικές κυβερνήσεις. Αν δεν γίνεται αυτό, έτσι δεν είναι. Ε, θα ήταν ιστορικά μοναδικό κάτι τέτοιο αν δεν το κάναμε τώρα. Δεν μπορώ όμως να προδικάσω τι θα πει η Επιτροπή Αλίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό ε, παρουσίασα το θέμα με αυτή τη μορφή της γνωμοδότησης. Εγώ υπολογίζω ότι θα αναβληθεί το θέμα και ότι θα ξανά αργότερα. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Αυτό είναι το θέμα. Τι άλλο να προσθέσω. Είπατε να ψηφίσουμε κατά. Δεν ξέρω αν είναι το σωστό αυτό, γιατί είναι η πρώτη μου θητεία στο Κοινοβούλιο και δεν ξέρω ακριβώς. Η Επιτροπή Αλληλείας είναι η αρμόδια επί της ουσίας. Αν συνεννοηθείτε να γίνει κάτι τέτοιο και να συμφωνήσουν όλοι. Δεν έχει σημασία αν θα γνωμοδοτήσουμε ή όχι. Γι' αυτό είπα, σε περίπτωση που θα γίνουν διαπραγματεύσεις να ψηφίσουμε ναι, γιατί για τη Γουλινέα Μπισάου είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία, δηλαδή αποτελεί ζωτική κριτικό παράγοντα για τη ζωή των ανθρώπων στη χώρα αυτή και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά να πούμε ότι αυτά τα αιτήματα έχουμε να διατυπώσουμε προς την Επιτροπή για την πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι δεν θα σκεφτεί. Ε, Ευχαριστώ όλους και όλες για τις ε, παρεμβάσεις σας συνθήκας. Θυμίζω τώρα η καταθέση τροπολογιών είναι η 13η Νοεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι, 13 Νοεμβρίου. Και συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το πολύ σημαντικό ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Πώς θα ανοίξουμε τον δρόμο πώς θα ξανανοίξουμε τον δρόμο στη βιώσιμη ανάκαμψη χωρίς υποκλεισμούς. Η Κατρίν Γκρέσ μου ζητά να εκφράσω τη λήψη γιατί απουσιάζει και μου ζήτησε να παρουσιάσω τα βασικά της γνωμοδότησής της. Κυρία Γκρέσ, λοιπόν, επιμένει επί δύο σημείων. Λέει ότι πρώτον, πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο από την εθελοντική προσέγγιση και να θεσπίσουμε νόμους, κανόνες δεσμευτικούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να αυτορυθμιστούν τη δική του μόνο πρωτοβουλία δεν οδηγεί πουθενά. Το βλέπουμε ε, στο τραπεζικό τομέα στι αναπτυγμένε χώρε, στην εξωτερική βιομηχανία στι αναπτυσσόμενε χώρε και στην Αφρική που ήμουν. Είδα ότι και εκεί δεν υπάρχει αντισυμβασμό για το περιβάλλον, ε, δεν πλέον φόρου αυτέ τι επιχειρήσει, δεν πληρώνουν εισφορέ, ε, δεν υπάρχει συμβασμό για τα δικαιώματα. Συνεπώ, το να είναι υπεύθυνη μητρική εταιρεία για τις ε, θηγατρικέ που ενεργούν σε αναπτυσμένες χώρες, αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Δείτε τι γίνεται για παράδειγμα στην Νιγηρία. Δείτε την στέρηση και την καταστροφή στο Δέλτα του Νίγηρα, όπου η παιδική θνησιμότητα είναι υψηλότερη σήμερα σε σύγκριση με πριν από 30 χρόνια. Είναι εύκολο να δει κανείς ότι το να αφήσει τις πολυεθνικές ελεύθερες να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς με δική τους μόνο πρωτοβουλία και κατά την κρίση τους δεν οδηγεί πουθενά. Στην Νότια είχαμε τα δραματικά περιστατικά τα πρόσφατα περιστατικά που μας ε, θυμίσουν ότι δεν γίνεται σεβαστό καν το δικαίωμα στην απεργία. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέους δεσμευτικού κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι μητρικές είναι υπεύθυνες για τη συμπεριφορά των θηγατρικών τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό πρέπει να θεσπίσουμε και δει για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με νέες οδηγίες. Επιπλέον, χρειαζόμαστε ένα σύστημα ελέγχου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις ε, επιχειρήσεις να επελθεύουν μόνες τους τις επιδόσεις τους. Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι στη, είτε στην Αμερική, είτε στην Ευρώπη, είτε στον αναπτυσσομενό κόσμο. Πρέπει λοιπόν να προσδώσουμε μεγαλύτερη λογοδοσία στο σύστημα. Έχουν συμβεί φοβερά πράγματα. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να θυμίσω τον Ήγηρα, που η Ερεβά, η γαλλική εταιρεία, η οποία εξάγει ουράνιο, μόλυνε την πηγή νερού για τους ε, αυτόχθονες πληθυσμούς. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι ακριβώς το αντίθετο. Αλλά αυτό ισχύει ως τώρα. Ανεξέλεγκτη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους χωρίς κανέναν έλεγχο ή καμία επιτήρηση. Αυτό ακριβώς πρέπει να, αλλάξουμε. Και αυτό είναι και το κεντρικό νόημα, η κεντρική ιδέα της ε, νομοδότησης της κυρίας Γκρέσ. Η Επιτροπή Επασχόληση είναι αρμόδια όπως και η Γιούρη, εμείς γνωμοδοτούμε. Πιστεύω ότι αυτά πρέπει να πούμε με την γνωμοδότησή μας. Να ζητήσουμε λοιπόν στην έκθεση αυτών των δύο επιτροπών να περιληφθούν τα στοιχεία τα οποία μόλις ανέφερα. Κύριε Κιόρεντς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κρέσ, ευχαριστώ μας είπατε έδειξε το ζήτημα, την καρδιά του ζητήματο και την ρίζα του. Συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Όμω, για να δούμε πρώτα τι πρόοδοι έχουν σημειωθεί στην διακυβέρνηση στις χώρες όπου επιχειρούν αυτές οι επιχειρήσεις. Απόλυτος απαραίτητο. Δηλαδή, αν μια χώρα έχει θεσπίσει αυστηρά πρότυπα για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, για, την, για για παράδειγμα, καλώς. Εδώ, στο πλαίσιο μιας άκροας ε, πριν με εκπρόσωπο της Νιγηρίας, ο οποίος μας είπε ότι για την εκμετάλλευση της χώρας του δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πλήρης αποτυχία, κυβέρνησης. Σπάνια έχω ακούσει τέτοια δήλωση, ομολογία εκ μέρους ενός καθεστώτος. Η συνεργασία μας λοιπόν με τις αναπτυσμένες χώρες πρέπει να συνεχίσει να ευνοεί την συγκεκριμένη πτυχή. Δεύτερον, ξέρουμε ότι στον τομέα αυτών τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αργά. Πρώτον, λόγω του ανταγωνισμού. Στον ΠΟΕ οι κανόνες είναι για όλους. Ξέρουμε όμως ότι η Κίνα με τις ε, πρακτικές εξασφάλισης πρόσβασης σε φυσικούς πόρους δεν μας επιτρέπει να ξέρουμε αν πληρώνει αρκετά, λιγότερο ή περισσότερο. Και πώς αξιοποιεί, ε, ενδεχομένω εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους που υποτίθεται ότι αξιοποιεί στο επίπεδο του ΟΣΑ και των, του ΟΗΕ υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο ΟΗΕ υιοθετεί το Παγκόσμιο Σύμφωνο, Global Compact. Καταγράφει λοιπόν τις δράσεις επιχειρήσεων που έχουν δραστηριότητες στο εξωτερικό. Εδώ μιλάμε για έναν κώδικα δαντολογίας, ο οποίος υποχρεώνει τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τέτοιου δραστηριότητες να δημοσιεύουν ετησίως τις πρόοδους που σημειώνουν σε δύο-τρεις τομείς. Και εδώ τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, είναι έως και αποκαρδιωτικά θα λέγα. Και τέταρτον, στο βαθμό που θέλουμε να είμαστε αυστηροί και να επιβάλλουμε έναν κώδικα δεντολογίας αλλά και κάτι περισσότερο, να επιβάλλουμε δηλαδή την τήρηση νομικών υποχρεώσεων, δεσμευτικών υποχρεώσεων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εγώ λέω ναι, Συμφωνώ, πρέπει να το πράξουμε, όμως προκειμένου πρέπει να εμπνευστούμε από αυτά τα οποία γίνονται εδώ. Α πούμε, εφαρμόζουμε την αρχή ορυπαίνων πληρών, γιατί να μην εφαρμοστεί, να μην ισχύσει για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα, για τις επιχειρήσει, που έχουν πρότυπα για την Ευρώπη, θα λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε τα ίδια πρότυπα και στο εξωτερικό. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι ηθικό μας καθήκον, ούτως ή άλλως, πέρα από το καθήκον μας προς το περιβάλλον. Κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσατε τις ιδέες ε, της συναδέλφου ε, κυρίας Γκρές είναι απόλυτα σωστός. Συμφωνώ απολύτως από το α μέχρι το ω. Τώρα το θέμα είναι πώς θα αναπτύξει η συνάδελφος κυρία Γκρέτς τις ιδέες αυτές στη συνέχεια στο κείμενο. Τη γνωρίζω βέβαια και γι' αυτό τρέφω πλήρη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της. Θα συντάξει το κείμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε όλοι επ' αυτού. Ο κύριος Γκέρενς πάντοτε διακατέχεται από κοινή λογική, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και δίνει τη δική του αποχρώσια έννοια σε ορισμένες διαστάσεις του θέματος. Ωστόσο, οι πολυεθνικές ή και μη πολυεθνικές επιχειρήσεις γιατί μπορούμε να, έχουμε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες να μην είναι πολυεθνικές και να δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν την ίδια νοοτροπία που έχουν και στην Ευρώπη. Δηλαδή στόχος τους είναι η μεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους τους. Και στην Ευρώπη σε κάποιο βαθμό έχουμε καταφέρει, σε κάθε πιο βαθμό λέω, αυτό το περιθώριο κέρδους να το ε, επιτρέπουμε μόνο υπό τον όρο ότι θα πληρούνται ορισμένες κοινωνικές προϋποθέσεις ή εργασιακές αν θέλετε προς υποθέσεις. Αλλά ε, αυτό το πράγμα για να το καταφέρουμε στην Ευρώπη χρειαστήκαμε δεκαετίες συνδικαλιστικής δράσης, ε, δράσης πολιτικής και άλλων ειδών, εν πάση περιπτώσει. Οι επιχειρήσεις όμως πάντοτε είναι ένα βήμα μπροστά και συνήθως κοροϊδεύουν, γελιοποιούν τους κανονιστικούς, ε, τις κανονιστικές διατάξεις και ρυθμίσεις που εγκρίνονται. Και είναι προφανές ότι κάθε φορά που έχουμε μια κανονιστική ρύθμιση πρέπει να γίνονται ε, περικοπές στο περιθώριο κέρδους. Τώρα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι διτό. Όσο περισσότερο ελέγχουμε και επιβάλλουμε κανόνες και διατάξεις στην Ευρώπη τόσο περισσότερο οι πολιεθνικές ή μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για να μην μιλήσω για τις βορειοαμερικάνικες, τόσο περισσότερο φεύγουν από την Ευρώπη και πάνε στις αναπτυσσόμενες χώρες για να έχουν τα περιθώρια κέρδους τα οποία δεν τους επιτρέπεται πλέον να έχουν στην Ευρώπη διότι πρέπει να εκπληρώσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε επίπεδο εργασιακού δικαίου ή περιβαλλοντικού δικαίου. Επομένως, οι εταιρείε αυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αυτά τα κέρδη διότι μπορούν να διαφύγουν από τους κανόνες και τους ελέγχους που εμείς καταφέραμε να θεσμοθετήσουμε στην Ευρώπη και αυτός είναι και ο μόνος λόγος για τον οποίο έχουν τόσο μεγάλα κέρδη. Από τη μία είναι αναξιοπρεπές να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο στον αναπτυσσόμενο κόσμο και από την άλλη αποτελούν πολύ σημαντικό ε, σημείο και στοιχείο ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία μετεγκατάστασης. Φεύγουν από την Ήπειρό μας, όχι γιατί δεν τους αρέσει το τοπίο ή δεν τους αρέσουν οι εργαζόμενοι, αλλά γιατί τους μειώθηκε αρκετά ο κέρδους ακριβώς λόγω των προϋποθέσεων που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή ε, Ήπειρο ε, ως προς τους περιβαλλοντικούς ή εργασιακούς όρους γενικότερα. Επομένως, και υπ' αυτή την έννοια, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκέρενς, το πρόβλημα είναι πώς θα καταφέρουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες να επιβληθούν παρόμοιοι όροι με αυτούς που καταφέραμε εμείς να επιβάλλουμε στην Ευρώπη. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που αναφέρει η κυρία Γκρές είναι ο έλεγχος. Και ο έλεγχος είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την έννοια της ευθύνης στην Ευρώπη είδαμε ότι σαφέστατα όταν οι επιχειρήσεις ε, αναλαμβάνουν την υποχρέωση αυτοελέγχου, αυτοελέγχονται μόνο και μόνο για να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους και όχι για να ε, ελέγξουν πραγματικά την συμμόρφωση με τους εργασιακούς ή περιβαλλοντικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα ήταν ιδιαίτερα ακριβό ε, η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων. Όμως, η ελεκτική δυνατότητα είναι μηδέν στις χώρες αυτές, για διάφορους λόγους. Και αυτό το παράδειγμα φαίνεται ε, ξεκάθαρα με την ε, εκμετάλλευση πετρελαϊκών, κοιτασμάτων σε μια χώρα την οποία δεν θα ονομάσω. Μια μικρή χώρα με πάρα πολλά κοιτάσματα. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε καμία δυνατότητα να ξέρουμε εάν αυτή τη στιγμή εξεωρίσετε, γίνεται γεώτρηση πετρελαίου με 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ή με 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Και δεν, δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί δεν υπάρχει κανένα έλεγχο, κανένα μηχανισμό ελέγχου. Ό,τι μα λέει ο πρόεδρο τη πολυεθνική θα πρέπει να το πιστέψουμε. Άρα, οφείλουμε να θεσμοθετήσουμε πλαίσια ελέγχου. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε στελέχη και μόλις τα εκπαιδεύουμε, τελικά τα στρατολογούν οι επιχειρήσεις και τους πληρώνουν 10 φορές πάνω από ό,τι εμείς. Αν εμείς τους δίνουμε 1000 ευρώ, ε, τον επόμενο μήνα τον προσλαμβάνει αυτό το στέλεχος κάποια επιχείρηση με μισθό 10.000 ευρώ. Επομένως, ε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει ελεγκτής με εκπαίδευση μετά προσλαμβάνεται και κάνει τον αυτοέλεγχο από πλευρά της επιχείρησης. Εξού και προσκρούμε σε τείχος. Ε, είναι σαφέστατες δηλαδή οι αρχές, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα. Ως Ευρώπη λοιπόν πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πρώτον, να διατηρήσουμε τους δικούς μας όρους και προϋποθέσεις και να τους βελτιώσουμε μάλιστα ε, τις προϋποθέσεις ως προς τους κανόνες και τους ελέγχους και από την άλλη να προσπαθήσουμε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, εν πάση περιπτώσει να μην είναι αυτές οι οποίες ε, ε, σε άλλες γωνιές του κόσμου ε, γελιοποιούν στο μεγαλύτερο βαθμό την, τις κανονιστικές διατάξεις που έχουμε εμείς σε ισχύ. Είναι ένας τρόπος αυτός να δράσουμε. Γιατί δεν προχωρούμε ε, πολύ σε διαφορετική περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι αξιέπαινες οι προσπάθειες της κυρίας Κρέζ, όπως και ε, οι προσπάθειες της συναδέλφου κυρίας Χόουιτ και του κυρίου Μπαλτασάβε. Ωστόσο, δεν παρετούμε δεν θέλω ε, να, έχω ητοπάθεια, αλλά επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στον τομέα αυτό, δεν ξέρω πραγματικά κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε πραγματική πρόοδο. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπέρ της ε, μη δράσης αλλά πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τις πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πόσο εμποδιζόμαστε σε αυτό το περίπλοκο εγχείρημα. Διότι αυτό το οποίο ισχύει και λέμε για τις αναψώμενες χώρες, πολύ συχνά ισχύει και μπορεί να ισχύει στις δικές μας χώρες μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βένσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέζ για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για την εταιρική και κοινωνική ευθύνη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όλοι εδώ συμφωνούμε πάνω στο εξής. Οι εταιρείε έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνη για την ανάπτυξη στις μικρές χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όντως μπορούν να επηρεάσουν ε, την ανάπτυξη και θα πρέπει αυτό να οδηγήσει και σε κοινωνική ανάπτυξη. Οι αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προέκυψαν ως αντίδραση στο γεγονός ότι ορισμένες επιχειρήσεις έδωσαν την πρωτοκαθεδρία στα βραχυπρόθεσμα κέρδη έναντι οποιοδήποτε άλλου τιμήματος ε, και η δραστηριότητα ήταν επικίνδυνη για τους εργαζομένους και επικίνδυνη και για το περιβάλλον. Επομένως, προέκυψαν οι αρχές κοινωνικής εταιρικής ευθύνης για να υπάρξει πρόληψη, να μην υπάρξει βλάβη από πλευράς επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων τους. Πρέπει όμως να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Δεν αρκεί αυτό που κάνουμε απλά να μην προκαλούν ζημία ή βλάβη οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι και ευεργετικές για την εκάστοτε χώρα, ότι κάνουν και καλό μάλιστα. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάλαβαν πόσα ωφέλη και οικονομικά και κοινωνικά ε, μπορούν να αποκομίσουν από τις αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οφείλουμε να ενημερώνουμε περισσότερο τους ε, καταναλωτές. Οι πολίτες, οι καταναλωτές είναι όλο και πιο ενημερωμένοι και περιμένουν τα τρόφιμα και όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν να έχουν παραχθεί με αηφόρο και υπεύθυνο τρόπο. Η καλύτερη το καλύτερο κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να ανεβάσουν τον πύχη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι η δύναμη των καταναλωτών, οι ενημερωμένοι καταναλωτές. Ε, αυτό είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό ε, με προβληματίζουν κάποιες διατυπώσεις στη γνωμοδότηση αυτή για τις νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις για τις ξένες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες π.χ. Ε, πολλές επιχειρήσεις έχουν καταλάβει ότι μακροπρόθεσμα θα χάσουν εάν δεν αναλαμβούν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ευθύνες βραχυπρόθεσμα. Εμένα η ένσταση μου ως προς ε, ε, τις υποχρεωτικές διατάξεις έχει να κάνει με, την, ε, το προσωρινό χαρακτήρα. Π.χ. στην εξορεκτική βιομηχανία έχουμε πάρα πολλές ε, παραβάσεις ε, της νομοθεσίας και όχι μόνο στην Αφρική αλλά και αλλού. Ενδεχομένως για αυτό το κλάδο της ε, οικονομίας, την εξορρυκτική βιομηχανία, χρειαζόμαστε ειδική εργαλειοθήκη, ειδικά μέσα δηλαδή στη διάθεσή μας. Βεβαίως θα υποβληθούν τροπολογίες, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Κρές και την ευχαριστώ για αυτό. δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί η κυρία Σουσεν Πάτ. Παρακαλώ. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Κομισιόν. Καλό σας απόγευμα. Να πω καταρχήν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρθησε ανακοίνωση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το CSR, τέλος του 2011, για να καλύψει αριθμό θεμάτων που δεν θα αναφέρω λεπτομερώς σήμερα, γιατί η έμφαση τώρα είναι η διεθνής πτυχή του CSR. Καλύπτει όμως την υποβολή εκθέσεων για τις ε, δραστηριότητες ε, από τις επιχειρήσεις, ε, εκπαίδευση, κατάρτιση στο CSR, δράσεις για την ορατότητα του CSR, την εμπιστοσύνη στις εταιρείε που θα το κάνουν, ε, επιβράβευση από την αγορά των εταιριών που κάνουν CSR. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης της Κομισιόν είναι αυτό που καλύπτει τα διεθνή θέματα και καλύπτει σχέσεις με άλλους διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, θεσμικά όργανα που ενδιαφέρονται για το CSR, όπως όσα οι κατευθυντήριες του όσα πολυεθνικές και το UN Global Compact, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ. Επίσης, για επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει ένα κομμάτι, ένα άλλο κομμάτι αφορά το, την αναπτυξιακή και εμπορική ατζέντα. Εμπόριο ανάπτυξη πάνε μαζί εκεί, με στόχο να προαχθούν οι επενδύσεις που θα είναι βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς για την προώθηση ναι. Οικονομικές, ε, ε, να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στις τρίτες χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή είναι η εισαγωγή για τις πολιτικές μας μέχρι σήμερα ή το πεδίο εφαρμογή και το σημείο όπου τα εφαρμόσαμε όλα αυτά μέχρι το τέλος της ε, περασμένης χρονιάς. Υπάρχει και η συνάντηση από την DG που συνεργασίας, ο γενικός στόχος της, των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης ε, βάσει συνθήκες της Λισαβόνας είναι η εξάλληψη της ε, φτώχειας. Το CSR είναι ένας τρόπος συνεργασίας με το ιδιωτικό τομέα για βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και ε, μείωση της φτώχειας. Η DG ε, ε, παρουσίασε μια ανακοίνωση για την αναπτυξιακή πολιτική και την ατζέντα για την αλλαγή. Τα ξέρετε αυτά που αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην πρόθεση της καινοτομίας, ε, την δημιουργία θέσεων την κινητοποίηση πόρων και τη συμβολή στον πολιτικό διάλογο. Η αλλαγή σε ενθαρρύνει εταιρικέ σχέσει συμπράξει μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου δομέα αναδεικνύοντα τη CSR και σε εθνικό και σε διεθνέ επίπεδο ω προ... μέσο προώθηση μια συμπεριφορά που συνάδει με διεθνώ αναγνωρισμένα πρότυπα και μέσα. Η ΤΕΦΚΟ επίση αναγνωρίζει ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα που στοχεύουν στι ανάγκε των φτωχών μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Ο ιδιωτικός τομέας παίζει μεγάλο ρόλο γιατί ε, δημιουργεί καλές υποδομές στην ενέργεια, στις ε, τεχνολογίες επικοινωνίας, ε, στην στέγη, στα φάρμακα και σε άλλους τομείς που διευκολύνουν και κάνουν καλύτερη τη ζωή των φτωχών ανθρώπων. Επίσης ε, εξετάζει την, τον αναπτυξιακό αντίκτυπο ε, όλων αυτών των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και που δίνουν καλά αποτελέσματα για αυτούς στη βάση της πυραμίδας. Θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε υποφελούνται οι φτωχοί όχι μόνο καταναλωτές, αλλά πιο σημαντικό ή εξίσου σημαντικό, δίνοντάς τους τα στοιχεία που χρειάζονται τους συντελεστές για τη δική τους την παραγωγή, ε, όπως ε, τους ε, μικρούς επιχειρηματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, τους αγρότες. Η DigiDevco διερευνά δυνατότητες για να διευκολύνει ανταλλαγή απόψεων και βελτίστων πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών εταιριών και να διεγείρει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υφισταμένων προγραμμάτων στήριξη από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ως πρώτο βήμα ανέθεσα μια μεγάλη μελέτη για την καλύτερη κατανόηση του τοπίου των προγραμμάτων σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα διαφόρων φορέων και για να δουν πού μπορεί να προσθέσει αξία σε αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας, Τώρα η Κομισιόν έλαβε υπόψη της τις ανησυχίες και μελήματα που υπάρχουν από τη συνεργασία για την ανάπτυξη με τις αναπτυσσόμενες χώρες και από τους εμπλεκομένους στην ατζέντα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Μέχρι τις 12 η το μεσημέρι 20 Νοεμβρίου έχετε χρόνο να υποβάλλετε η ψηφορία 6 Δεκεμβρίου. Και περνάμε στο 11ο σημείο της σημερινής διάταξης πρόθεση ανάπτυξης μέσω εμπορίου. Εισηγητής ο κύριος Σβένσον. Παρακαλώ κύριε Σβένσον. Πρόεδρε, εισαγωγικός να θυμίσω πώς φτάσαμε στην έκθεση. Αυτή είναι μόνο η μισή απάντηση, θέλετε, στην πρωτοβουλία του Επιτροπού Ντεχούχτ. Να βοηθήσουμε τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο την βοήθειά μας. Ξεκίνησε με 27 Ιανουαρίου έχει περάσει τον ένα χρόνο από τότε. Και ξαναλέω ότι είναι η μισή μα απάντηση, η μισή ανταπόκριση του Κοινοβουλίου και του διότι η κυρία Τόκια Σαϊφή του ΕΛΚ αυτήν την στιγμή συγγράφει μια άλλη έκθεση στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Το Κοινοβούλιο λοιπόν δεν έχει ακόμη αποφανθεί και τούτο διότι να το θέσω διπλωματικά, υπήρχε μια ευγενή άμυλα μεταξύ των δύο επιτροπών για το ποιο θα υποβάλει έκθεση. Είναι τα ΙΝΤΕΒΕ. Βεβαίω, καταρχήν είναι επίτροπο για το εξωτερικό εμπόριο. Έλαβε την πρωτοβουλία, άρα προηγείται κατά κάποιο τρόπο η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Όμω, και εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή μα ε, είναι αρμόδια ή τουλάχιστον εξίσου σημαντική ω προ το θέμα αυτό. Ξέρω ότι οι σχετικέ διαπραγματεύσει μεταξύ των επιτροπών κράτησαν αρκετά και καταλήξαμε σε μια σαφή διάκριση των αρμοδιοτήτων μας. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι θα συνταχθεί μια έκθεση και ότι θα αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Αν λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρείτε ότι στο έγγραφο εργασία το οποίο έχουμε μπροστά μα λείπει μία ή η άλλη άποψη, οπτική γωνία, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονό ότι η κατανομή εργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μπορεί να ε, σημαίνει ότι η κυρία Σάιφη έχει αναλάβει αυτέ τι πτυχέ να τι καλύψει. Να ευχαριστώ λοιπόν του φίλου από την γραμματεία τη ΤΕΒΕ, οι οποίοι έλαβαν μέρο στι διαπραγματεύσει μεταξύ των δύο επιτροπών πραγματικά έδωσαν σκληρή μάχη με νύχια και με δόντια για να εξασφαλίσουμε ότι περισσότερο μπορούμε. Οπότε, τώρα που τελείωσαν αυτά, ας δούμε τις λεπτομέρειες. Να σας πω τώρα την δική μου άποψη για τη συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη στις φτωχές χώρες. Όπως ε, λέω και στο κείμενο, είμαι πεπισμένος ότι το εμπόριο είναι ο κατεξοχήν τομέα στον οποίο μπορούμε να αποδείξουμε την συνοχή των παρεμβάσεων μας. Τα πολιτικά αυτά εργαλεία στον τομέα του εμπορίου μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη στις φτωχές χώρες περισσότερο από ότι οι καθευτό αναπτυξιακές πολιτικές. Το εμπόριο πρέπει να υποστηρίζει τις προτεραιότητές μας στον τομέα της ανάπτυξης. Αυτό λέγεται βεβαίω στην ανακοίνωση της Κομισιόν, αλλά εμπαρόδο θα μπορούσε να γίνει πιο έντονο. Για παράδειγμα δεν γίνεται κανένα σχολιασμό στην αξία των διαφόρων μορφών εμπορίου και το πώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη και πώς αυτή η συμβολή μπορεί να μεγιστοποιηθεί. Επίσης, εν παραδόκι μόνο, αναφέρεται το ότι το εμπόριο μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις επί των αναπτυσσομένων χωρών. Γι' αυτό εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα ζητήματα αυτά για να διασφαλίζουμε ότι θετική ανάπτυξη μπορεί να προκληθεί από το εμπόριο. Και ότι όλα αυτά μπορούν να μεταφραστούν σε κοινωνική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη χωρί δικαιώματα του ανθρώπου, για παράδειγμα, χωρί πολιτικέ ελευθερίε, δεν έχει πολύ νόημα. Η δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι εκτρονοκάνευ για την αηφόρο ανάπτυξη μια χώρα. Γι' αυτό και η πολιτική, η εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκής Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προβλέπει και συγκεκριμένους στόχους και να διασφαλίζει ότι όλα αυτά όντω γίνονται σεβαστά. Ο έλεγχο δηλαδή για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου πρέπει να ενσωματώνεται στου μηχανισμού μα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το εμπόριο με τι αναπτυσσόμενε χώρε να εκδηλωθεί ω άσκηση υπεροχή επί των πλέον αδυνάτων. Όχι, πρέπει να είναι μια ισότιμη σχέση με τι φτωχότερε χώρε. Επίση, δεν πρέπει να πρόκειται περί προστατευτισμού αντί ημών ή άλλων χωρών. Οι συμφωνίες εμπορικέ με τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να προβλέπουν και δικές μας θυσίες, όχι μόνο από την άλλη πλευρά. Στην έκθεση αυτή καθ' αυτή φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτούς τους λογισμούς περαιτέρω, πέρα από το έγγραφο δηλαδή εργασίας να πούμε ακριβώς πώς βλέπουμε το εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και δει τα μέτρα που μπορούν να αποβούν χρήσιμα. Κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω και το οποίο θεωρώ χρήσιμο είναι το εξή. Υπάρχει μεγάλη ηθική και περιβαλλοντική ευθύνη για την ευρωπαϊκή Ένωση. Και δει για την εξωτερική βιομηχανία στι αναπτυσσόμενε χώρε. Το είπαμε αυτό προηγουμένω. Αυτό αφορά όχι μόνο τι διεθνεί εταιρείε, τι πολυεθνικέ, αλλά και τι εγχώριε που δραστηριοποιούνται στην εξόριξη. Προσβλέπω στην ανταλλαγή υπόψεων με του ε, συναδέλφου. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη φιλοδοξή έκθεση, η οποία θα είναι υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών οι οποίε έτσι θα υποφεληθούν από το διεθνέ εμπόριο. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Νόησα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Σβένσον για την καλή συμβολή στο θέμα εμπόριο και ανάπτυξη η διευκρίνηση ήταν επίσης σημαντική ότι εμείς ως μέλη στην Επιτροπή Ανάπτυξης θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τη θεματική αυτή όσο γίνεται περισσότερο. Να μην τα αφήσουμε μόνο στην Επιτροπή Εμπορίου. Για την ομάδα μας, κύριε Σβένσον, μπορώ να πω ότι συμφωνούμε με τις θέσεις σας Πολλούς σημαντικούς τομείς ε, αναφέρατε από το θέμα εμπόριο και ανάπτυξη και η θέση αυτή νομίζω ότι θα αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση αργότερα. Θέλω να αναφερθώ σε κάποια βασικά θέματα, πολύ βασικά για μας. Δυστυχώς ε, το εμπόριο και η οικονομική ανάπτυξη δεν ανταποκρίνονται πάντοτε, δεν μεταφράζονται πάντοτε σε θετική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό βέβαια και η οικονομία και το εμπόριο να ανακάμπτουν, αλλά αυτό δεν αρκεί για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής ε, των, ε, του κόσμου στον, ε, στις χώρες εταίρους. Θα πρέπει η, το εμπόριο και η οικονομική ανάπτυξη να επιδρούν στην ανάπτυξη θετικά και θα πρέπει το εμπόριο να συνδυάζεται με ευφυή πολιτική. Καλή διακυβέρνηση. Μιλήσατε για τις ευρωπαϊκές βασικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα και που θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη στις εμπορικές συμφωνίες και τα περιβαλλοντικά στάνταρ προσθέτω εγώ, τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Πιστεύουμε ότι το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ο ILO, με το πρόγραμμα των κοινωνικών ελάχιστων προτύπων, έθεσε καλές βάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να υποστηριχθούν. Καταρχήν, το εμπόριο οδηγεί σε περισσότερη εργασία και περισσότερες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και με, που ξεπερνά την εξαγωγή πρώτων υλών. Η εμπορική βοήθεια, το Aid for Trade, είναι πολύ σημαντική για μας. Εδώ συγκαταλέγεται η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση των φορολογικών και δημοσιονομικών συστημάτων των χωρών εταίρων μας, ούτω ώστε να ενισχύεται το σκέλος των εσόδων. Πρέπει να ε, εμποδίσουμε η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική να οδηγήσει σε φορολογικό και κοινωνικό dumping. Μια τελευταία λέξη ακόμη για τις διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών. Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βένσον, θα πρέπει να ε, είναι ε, ορατές, ε, ε, εύληπτες και θα πρέπει να υπάρχει και εκπαίδευση και κατάρτιση στα Υπουργεία Εμπορίου των χωρών εταίρων μας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εξάρτηση από το εξωτερικό, θα πρέπει και εκείνοι με τρόπο επαγγελματικό να προασπίζουν τα συμφέροντά τους και σε διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες και με άλλα κράτη αυτό θα τους χρησιμεύσει πολύ. Είναι καλή βάση αυτή ε, που μας δώσατε και νομίζω ότι πολύ γρήγορα τις επόμενες εβδομάδες μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκιόρεντς. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι το 10 και 11 θα μπορούσαμε να τα συγκεράσουμε και να τα ζητήσουμε μαζί. Τα ζητήματα είναι ομοίδη, συνδέονται μεταξύ τους. Τώρα ως προς το εμπόριο ως μέσο αύξηση του πλούτου όλοι συμφωνούμε το γνωρίζουμε αυτό, συμφωνούμε με τη δεύτερη διαπίστωση όταν δημιουργείται πλούτος προφανώς δεν ε, δημιουργάζεται αυτομάτως δίκαια. Ο στόχος είναι εκείνος Βεβαίω θέλουμε να εξαλείψουμε την φτώχεια, αλλά δεν έχουμε τα μέσα για να επιβάλλουμε ακριβώ την καλή κατανομή του πλούτου, ο οποίο δημιουργείται στι αναπτυσσόμενε χώρε. Αν κατάλαβα καλά, το κείμενο αυτό θα γίνει ψήφισμα. Σε αυτό το ψήφισμα πρέπει οι συμπεφωνημένες μεταξύ μας αρχές να οδηγούν και σε λύσεις ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, που είναι αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Το είπαμε άλλωστε με την ευκαιρία της έκθεσης για τη μελλοντική ατζέντα της ανάπτυξης. Αυτό είναι μία αρχή. Αυτό μας το οποίο προσδοκούμε είναι να διαδερματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικότερο ρόλο για την εξάλληψη της φτώχειας. Χωρίς φυσικά αυτό να μπορούμε να το εγγυηθούμε. Κατά τα άλλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοείται ότι κάνει την πορεία στα διεθνή φόρα, ας πούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και στην Παγκόσμια Τράπεζα, που σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνα, αν όχι ε, συνυπεύθυνα για την διαμόρφωση των ενεργειών μας σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, Υπηρεσία για την Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να διαδραματίσει ε, σοβαρό ρόλο. Κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τη δουλειά του κυρίου Σβένσον. Είναι πολύ σημαντική. Και πολύ σημαντικό είναι επίσης ε, η δική μας Επιτροπή και όχι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου επιτέλους να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Αφού και οι δύο εισηγητές ανήκουν στην ίδια πολιτική ομάδα ε, και συμφωνούν γενικότερα, σίγουρα δεν θα υπάρχουν διαφωνίες. Όμως θα πρέπει να υπερασπιστούμε τις προτεραιότητες που έχει η δική μας Επιτροπή για διάφορους λόγους, αλλά και για τον εξής λόγο. τα θεσμικά όργανα και οι φορείς και ο κόσμος με τους οποίους ε, βρισκόμαστε εμείς σε καθημερινή επαφή είναι ακριβώς αυτοί που θα υπογράψουν αυτού του είδους τις συμφωνίες. Θα ήθελα να κάνω το εξή σχόλιο. Όπως ε, θα ξέρετε, την επόμενη χρονιά θα γίνει μια πολύ σημαντική σύνοδος μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ανέκαθεν, επί τη ευκαιρία των συνόδων, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν παρόν με ένα έγγραφο που παρουσίαζει την τοποθέτησή του. Θα πρέπει να πάμε πιο πέρα, να ξεπεράσουμε αυτές τις γενικότητες που λέγαμε σε ορισμένες από τις παλαιότερες συνόδους. Και νομίζω ότι στην έκθεση του κυρίου Σβένσον πράγματι υπάρχει περιεχόμενο, υπάρχει υλικό ώστε η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συναντηθεί με τα μέλη των Αφρικανικών Κοινοβουλίων ώστε να καταλήξουν σε ένα κοινό έγγραφο το οποίο θα παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής Αρχικών Κρατών και Κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής να καταλήξουν σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις εμείς και εμείς με ήττα και ύψιλον ώστε να υποβληθεί τελικά το έγγραφο αυτό στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτό είναι και το βασικό θέμα που θα συζητηθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το κείμενο του κυρίου Σβένσον για τις καθημερινές κοινοβουλευτικές μας εργασίες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μαγιά για να ε, καταλήξουμε στην τοποθέτησή μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Αφρικανικά Κοινοβούλια επίσης, ε, εν ώψη της επόμενης συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις γενικότητες που έχουμε εκφράσει στο παρελθόν, τις διάφορες συναντήσεις για λόγους πρωτοκόλου που έχουμε οργανώσει στο παρελθόν. Θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένα μέσα στη διάθεσή μας και αυτό είναι ένα πολύ ε, χρήσιμο και συγκεκριμένο μέσο, η έκθεση δηλαδή του κυρίου Σβένσον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, ένα ευχαριστώ στον κύριο Σφένσον για το εξαιρετικό έγγραφο εργασία. Θεμέλιο για το μέλλον. Θίξατε σημαντικά ζητήματα. Μεγάλη σημασία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για παράδειγμα, όντως το εμπόριο πρέπει να υποστηρίξει την πολιτική ανάπτυξης το εμπόριο δεν έχει και πολύ νόημα αν δεν συμβάλλει προς αυτόν τον στόχο. Λέτε επίσης ένα όχι στον προστατευτισμό, στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης τονίζετε τη σημασία μιας προσπάθειας η οποία θα ξεκινάει από τη βάση. Εξαιρετικό το κείμενο, πολύ το είπαν αυτό. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με βάση το κείμενο για να καταλήξουμε σε ένα άλλο εξαιρετικό κείμενο. Διαβάζοντα πάντως τις απόψεις αυτέ βλέπω ότι ξεχάσατε κάτι και θα ήθελα να το τονίσω. Το εμπόριο δεν είναι σκοπό. Όχι. Υπηρετεί άλλους σκοπούς. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Πρέπει να δούμε το εμπόριο, όχι βεβαίω ω ε, πανάκια, αλλά ως πολιτική η οποία μπορεί να λύσει ορισμένα προβλήματα. Δεν το λέτε έτσι ακριβώς, ίσως το υπονοείτε, αλλά θα ήθελα να το πούμε. Έχουμε ίσως εδώ την ευκαιρία να θυμίσουμε και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Πώς το εμπόριο δηλαδή μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της αηφορίας, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται του κλίματος. Κάτι άλλο επίση. η πτυχή που αφορά τα δύο φύλλα. Γυναίκε και άνδρες επηρεάζονται με πολύ διαφορετικού τρόπους στις αναπτυσσμένε χώρες από την ανάπτυξη. Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι τομεί που θα μπορούσαμε να αναδείξουμε εδώ, λαμβάνοντα υπόψη την πτυχή τη ισότητα. Εγώ υπόσχομαι από την πλευρά μου ότι θα συμβάλλω για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό κείμενο. Κύριε Σβένσον, και εγώ σας ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, για την εργασία σας που αποτελεί εξαιρετική βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Να τονίσω και εγώ κάποια από τα σχόλια της Κομισιόν, τα οποία μου φαίνεται ότι δεν ευνοούν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, με η Κομισιόν πολύ στις διμερείς διαπραγματεύσεις ή τις διαπραγματεύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Μια προσπάθεια που απέτυχε ακριβώς λόγω των δισταγμών των αναπτυσσομένων χωρών. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να κινηθούμε διμερός δεν σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να απελευθερώσουμε ακόμη περισσότερο το διμέρες εμπόριο. Τώρα, οι παρεμβάσεις του Δούνου του δείχνουν ότι όταν υποχρεώνουμε τις χώρες στο πλαίσιο της απελευθέρωσης να καταργήσουν δασμούς, για παράδειγμα είτε εισαγωγικού είτε εξαγωγικού, οι χώρες αυτές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα έσοδα αυτά με το ΦΠΑ. Μόνο ένα τρίτο μπορούν να υποκαταστήσουν. αυτό είναι δυστυχώ η πραγματικότητα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να αποστερήσουμε τις αναπτυσσόμενε χώρες από αυτό το εργαλείο και δι' τους εξαγωγικούς δασμούς. Για παράδειγμα, εξάγουν τεράστιες ποσότητες ε, χαλκού. Η επιβολή ενός ε, εξαγωγικού δεσμού δεν αποτελεί σημαντική γραφειοκρατία. Μια πολυεθνική έχει εξαιρετικό λογιστικό σύστημα, λίμωνο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα αυτό για την κατάργηση του εξαγωγικού δεσμού. Το ίδιο για τις άμεσε ξένες επενδύσεις. FDI. Το ότι αναπτύσσεται το εμπόριο, το ότι γίνονται επενδύσεις, δεν σημαίνει αυτομάτως και ωφέλη για τον τοπικό πληθυσμό. Φυσικά αυτός είναι ο στόχος. Αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος επί 40 χρόνια θα έλεγα δεν βλέπω να επιτυγχάνεται. Ένα απέσιο παράδειγμα είναι η Χιλίο που το αρχείο της Έξον δεν άφησε το παραμικρό κέρδος για τη χώρα επί 25 χρόνια. Μηδενικά κέρδη, μηδενικά ωφελήματα. Χρησιμοποίησαν τις υποδομές της χώρας, εκμεταλλεύτηκαν τον πλούτο της χώρας. Λοιπόν, βλέπετε ότι μία δραστηριότητα από μόνη της δεν, επαρκεί, δεν αρκεί για να έχει κέρδη η χώρα. Ας το πούμε λοιπόν αυτό. Οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη και έχουν, θα λέγα, καθήκον κάθε φορά που επενδύουν. Δεν είναι δικαίωμα. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Δεν αρκεί λοιπόν η Coca-Cola να μας εξηγεί στην ετήσια εκθέσή της ότι δημιουργεί δημιουργικά σχολεία για τους Ινδιάνους. Καλό αυτό, αλλά δεν μας λέει πόσα βαρέα μέταλλα, πόσες ε, φιάλες ε, άφησαν εδώ και εκεί και ποια ήταν η κατανάλωση του νερού στις περιοχές των Ινδιάνων. Θεωρώ λοιπόν, το ξαναλέω, ότι πρέπει να σχολιάσουμε τις απόψεις της Κομισιόν και να καταγράψουμε τη δική μας οπτική γωνία που κατατείνει στο ότι δεν αρκεί απελευθέρωση, χρειάζονται και ρήτρε προστασία, συνοδευτικά μέτρα ώστε να εξελιχθούν όλα όπω πρέπει. Και ξαναδίνω το λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Ντενί Μπαγέ. Um, thank you, um, Ε, την ε, εξωτερική και παγκόσμια διάσταση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένη η ανακοίνωση αυτή. Ενημερώνει την ανακοίνωση του 2002, συμπεριλαμβάνοντας τις νέες εξελίξεις. Πολλές πτυχές της προηγούμενης ε, ανακοίνωσης ισχύουν ακόμα και σήμερα. Σε 10 χρόνια όμως Κάθε δέκα χρόνια βεβαίως υπάρχουν αλλαγές, ο κόσμος είναι αλλαγμένο δέκα χρόνια πριν, σε σχέση με δέκα χρόνια πριν και γι' αυτό πρέπει να ενημερώσουμε την ανακοίνωση αυτή, εξού και το κάναμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθώ σε δύο βασικές πτυχές. Πρώτον, στο σχέδιο γνωμοδότησης, και να πω ότι εδώ δεν υπήρχαν πολλές διαφωνίες και μάλιστα μεγάλη σύγκληση είδα μεταξύ της ανακοίνωσης της δικής μας ως Ευρωπαϊκή, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, των παρεμβάσεων εδώ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να διευκρινίσω ορισμένα σημεία, εν συντομία. Πρώτον, ο βασικός στόχος ανακοίνωσης είναι ε, να είναι μια, πιο ενημερωμένη εκδοχή της ανακοίνωσης του 2002 και έχουμε και την ατζέντα για αλλαγή ως ε, υλικό Έχουμε τη συνένεση για τις αναπτυξιακές πολιτικές και το Aid for Trade, ε, το γνωστό. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της αναπτυσσόμενες χώρες και τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ως προς τις λεπτομέρειες ε, του σχεδίου κειμένου που έχετε μπροστά σας, ήδη εμπορίου. Πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν χρησιμοποιήσαμε πολλές λέξεις για να περιγράψουμε όλα τα δυνατά είδη εμπορίου. Θα ήταν όμως ενδεχομένως χρήσιμο να τα εξετάσουμε αυτά τα ίδια εμπόριο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο εισηγητής θέλει να μάθει περισσότερα π.χ. για το δίκαιο εμπόριο, για το αϊφόρο, το βιώσιμο εμπόριο. Καλό θα ήταν όμως να είμαστε σαφείς μεταξύ μας. Τι ε, θεωρείτε ότι λείπει από το κείμενο εδώ. Τώρα, ως προς τις ε, δυσμενείς επιπτώσεις ή τις ε, παρενέργειες, αν θέλετε, τις δυνατές. Πάντοτε στις μεταρρυθμίσεις υπάρχει αυτός ο φόβος. Κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Κανείς δεν είπε ότι η άμεση και πλήρη απελευθέρωση, άμεση και πλήρης απελευθέρωση είναι η μαγική συνταγή. Σε καμία ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λέγεται κάτι τέτοιο. Όλες οι κινήσεις πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες και θα πρέπει να προβλεφθούν τυχόν παρενέργειες και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να μην υπάρξουν τέτοιου είδους παρενέργειες. Τώρα, σε κάθε εμπορική συμφωνία έχουμε ρήτρε που αναφέρονται στο τόσο σημαντικό ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Σύμβαση Κοτονού βεβαίως και υπάρχουν τέτοιου είδους διατάξεις, αλλά και σε άλλα διμερεί εργαλεία. Γίνεται αναφορά και σε υψηλότερους δασμούς για τα μεταποιημένα προϊόντα σε σχέση με τις πρώτες ύλες. Ε, δεν είναι καινούριο επιχείρημα, ε, δεν έχει όμως και τόσο μεγάλη σχέση πλέον σε όλες τις χώρες αυτές, τις λιγότερο αντεπτυγμένες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει απαλλαγή από αλλά και σε άλλες. Άλλωστε είναι μια άτυπη, ένας άτυπος κανόνας του ΠΟΕ, ότι η απελευθέρωση πρέπει να φτάσει μέχρι και το 80%. Ε, σε κάθε περίπτωση το βάρος που έχει η δασμολογική πολιτική και η επιβολή δασμών είναι όλο και λιγότερο πλέον στο διεθνές στερέωμα, εκτός από πολύ συγκεκριμένου και λίγους τομείς της οικονομίας. Ως προς τις φήμες για τις πιέσεις που ασκούνται για την υπογραφή των συμφωνιών, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη αναφορά αυτή που γίνεται. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να υπογράψει μια συμφωνία που δεν θέλει να υπογράψει. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι ξέρει ότι αυτό έχει πράγματι συμβεί κάπου, ότι υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όλα τα ε, ε μέρη ε, το κάνουν ε, διότι έχουν αυτή τη βούληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δική της κόκκινη γραμμή. Υπάρχουν χώρες με, τους οποίους δεν θα, με τις οποίες δεν θα υπογράφαμε ποτέ συμφωνία, γιατί αυτό θα ήταν κατά ορισμένων κανόνων του ΠΟΕ ή γιατί οι χώρες αυτές ε, έχουν πολιτικές με τις οποίες διαφωνούμε καθέτας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί και να δούμε για ποιους λόγους έχουν κυκλοφορήσει τέτοιου είδους φήμες κάθε φορά που τις συναντούμε. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να πω και το εξής. Ε, με εξέπληξε κάπως η δική σας παρέμβαση. Η ανακοίνωση ρητός αναφέρει ότι οι, οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ είναι και η άγουσα που προτιμούμε αλλά θα πρέπει με ρεαλισμό να αποδεχθούμε την πολύ βραδία πρόοδο που σημειώνεται στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να εξετάσουμε και το εδεχόμενο να προχωρήσουμε γρηγορότερα ή πιο μακριά με ορισμένους από τους εταίρους οι οποίοι είναι έτοιμοι και επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε την μία οδό όταν επιλέγουμε την άλλη, εκεί όπου αυτό είναι σκόπιμο και εφικτό. Ως προς το φόρο επί των εξαγωγών η Κομισιόν ήταν πολύ ευέλικτη στις διαπραγματεύσεις αυτές. Πολλοί οικονομολόγοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι αυτό το εργαλείο δεν είναι και το βέλτιστο της επιστροφής του φόρου, δηλαδή κατά τις εξαγωγές. Είναι δύσκολο να εξαλειφθούν πλήρως ε, σταδιακά και είναι και αντικείμενο διαπραγματεύσεων θα ήταν επικίνδυνο η σύσταση να περιλαμβάνει ε, την υιοθέτηση ε, αυτού του είδους των ε, εξαγωγικών επιστροφών φόρου. Δεν θα έβρισκε σύμφωνος, σύμφωνη μεγάλη μερίδα των οικονομολόγων. Θα προτείναμε εμείς μια ισορροπημένη προσέγγιση. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι δεν ταυτίζουμε την απελευθέρωση με την ανάπτυξη. Αυτό που λέμε είναι ότι πολύ συχνά και υπό ορισμένε προϋποθέσεις ε, μια καλά σχεδιασμένη απελευθέρωση ε, ε, των αγορών μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση και είναι αυτό κάτι που αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Σβένσον. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος ως συνήθως κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλους όσους παρενέβησαν για τα ευγενικά σχόλια. Όπως είπα στην εισαγωγή, θα υπάρξουν κάποιες πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο από την ίντα. Θα δούμε τι θα πούν. Είναι διαφορετικές μορφές εμπορίου Μπορεί να είναι σε βασικά αγαθά, σε μεταποιημένα προϊόντα, σε πρώτες ύλε. Είναι σημαντικό όμως να υπογραμμίσουμε αυτό που λέγεται ότι σε πολιτικό επίπεδο το εμπόριο ε, από μόνο του δεν είναι εγγύηση ούτε για την οικονομική ανάπτυξη. Ε, ε, ε, η οικονομική ανάπτυξη πολλές φορές, θεωρείται αυτός σκοπός που και αυτός δεν είναι. Όπως είπαν ε, πολλοί συνάδελφοι σωστά, το εμπόριο πρέπει να συνδυάζεται με κάτι παραπάνω από συμφωνίες και διατυπώσεις, αλλά με απτά, ορατά ε, βήματα σε κοινωνικό επίπεδο που θα βοηθούν ελευθερίες και δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα θυμάστε ότι έχουμε αλλάξει την ημερήσια μας διάταξη. Δεν θα εξετάσουμε το σημείο 12 σήμερα. Θα το εξετάσουμε στις 6 Δεκεμβρίου, όπως ζήτησε ο εισηγητής κύριος Κάσμαν. Εξετάζουμε λοιπόν τώρα το σημείο 13 της ημερησίας διάταξης, ενδιάμεση συμφωνία η οποία θεσπίζει το πλαίσιο ε, μια συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της ε, ε, Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκίτρια είναι η κυρία Σαρτζεντίνη, η οποία δεν είναι εδώ και γι' αυτό την αντικαθιστά ο κύριος Μπαχτ Στάς, στον οποίο θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Τζούδη δεν μπόρεσε να έρθει και ζητεί συγγνώμη. Σύντομα, η αρχική ομάδα των χωρών της Ανατολικής ε, Αφρικής που αρχικά υπέγραψαν ήταν 16 χώρες. Δεν και είμαι αυθεντική ε, Αφρική. Τώρα 6 υπέγραψαν και 4, μάλλον 6 συνήψαν και 4 υπέγραψαν. Μαδαγασάρι, Μαυρίσιο, Σιχέλη, Ζιμπάμπου. Οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει και πολύ ενθουσιασμός για αυτά τα πράγματα. Ούτε αυτό είναι κομμάτι γνήσιας αναπτυξιακής ατζέντα σε, αυτά, σε αυτές τις προσωρινές ε, οικονομικές εταιρικές σχέσεις. Ε, υπάρχουν διαφορές ε, από χώρα σε χώρα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάργησης των δασμών και η κυρία Σαρτζεντίνη, το κείμενο των συμφωνιών είναι το ίδιο όμως, η κυρία Σαρτζεντίνη όμως στην αιτιολόγηση παρουσιάζει κάποια νούμερα που δείχνουν πόσο αρνητική θα είναι αυτή η συμφωνία για τις χώρες αυτές που θα σουν φορολογικά έσοδα, η Μαγαδαγασκάρη που είναι από τις λιγότερο αναπτυγμένες, λιγότερο λιγότερη αναπτυγμένη από τις τέσσερις, εκεί η συμφωνία είναι ακόμα λιγότερο υποφιλής από την τωρινή ρύθμιση που έχουν τη συμφωνία ΕΜΠΑ που είναι οτιδήποτε εκτός από όπλα είναι λιγότερο καλή από τις συμφωνίες ε, στα πλαίσια του Κοτονού. Ε, επίσης, η κυρία Σαρτζεντίνη στη σύντομη αιτιολόγησή της λέει ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη εδώ, ούτε ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και φαίνεται ότι η συμφωνία αυτή δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την περιφερειακή ολοκλήρωση λόγω σημαντικών διαφορών στην απελευθέρωση των δασμών ε, και τη διαδικασία κατάργησης των δασμών. Αυτό αφορά γιατί θα κάνουμε στο μέλλον. Αλλά δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι το Φεβρουάριο του 2009 υπήρξε ένα ψήφισμα όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια είπε ότι το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν να μην υπογραφούν αυτές οι οικονομικές ε, εταιρικέ ε, συμφωνίες γιατί συνιστούν προβλήματα και κινδύνους και η κυρία Αργεντίνη συμφωνεί με αυτή την άποψη και προτείνει η Επιτροπή μας να μην συγκατατεθεί ε, στις συμφωνίες αυτές και θα πάει αυτό στην Επιτροπή Ίντα που είναι και η Επιτροπή Αρμόδια επί της ουσίας. Ελπίζω να την εκπροσώπησα καλά την κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ να δώσω το λόγο στην κυρία Σνάιμπερ Γιάστραμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριο, κύριο Σβένσον, ο σκιώδης εισηγητής για αυτό το τομέα, έπρεπε να φύγει τώρα και να υποβάλει έκθεση μια άλλη επιτροπή. Με παρακάλεσε λοιπόν να σας πω τα κάτωθη. Ως εισηγητής ε, της ομάδας ΕΛΚ θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Σαρτζεντίνη για τη γνωμοδότησή της για τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Συμφωνώ με την κριτική της κυρίας Σαρτζεντίνη σε πολλά σημεία. Παρ' όλα αυτά είμαι βέβαιος ότι μια σύντομη ε, σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης εταιρικής σχέσης θα βοηθήσει τις χώρες και την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Γι' αυτό θα καταθέσω μια τροπολογία και παρακαλώ και συστήνω στο Κοινοβούλιο να ε, υπερψηφίσει αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μιλώ εξ του σκιώδους μας, του Μάικλ Κάσμαν και θέλω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν ευχαριστή για την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης της συμφωνίας. Η συμφωνία είναι κρίσιμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις χώρες ESA, Ανατολικής και Μεσημερικής Αφρικής. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ έντονες, όχι πολύ παραγωγικές όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρήκε τρόπους να υιοθετήσει, να συμβιβάσει ε, επιθετικές απόψεις και να παρουσιάσει ως γεγονός αυτές τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης της ΕΠΑΣ. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Μια παρατήρηση είναι ότι ενώ το βάρος της συμμόρφωσης ε, με τις ρήτρες συχνά ε, αφορά τόσο της, την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις χώρες ΑΚΕ, το κόστος προσαρμογής σε μεγάλο βαθμό ε, βαρύνει την πλευρά της τον χρόνο και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή ε, πιστεύουμε ότι οι συμφωνίες αυτές θα συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ και θα προάγουν, την ανάπτυξη ε, παράλληλα με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες των αντίστοιχων χωρών ΑΚΕ και τις περιφέρειες. Και οι δύο πλευρές των διαπραγματεύσεων, τα δύο μέρη έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη κάποιων επίμαχων θεμάτων μέσα στις συμφωνίες και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να δείξουν την προθυμία να εξετάσουν τα επίμαχα και εμφισβητούμενα θέματα και να υιοθετήσουν ευέλικτες προσεγγίσεις προς τα θέματα αυτά στα πλαίσια των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για πιο συνεκτικές ε, συμφωνίες. Ε, αυτή η μεταβατική συμφωνία μπορεί να το κάνει αυτό. Εμείς θα πρέπει να δούμε τι θέση θα ε, υιοθετήσουμε, θα εξετάσουμε δηλαδή στην ομάδα μας, γιατί το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, εξ όσων γνωρίζω, είναι υπέρ και άλλη επιτροπή μάλλον τάσεται κατά της έγκρισης του σχεδίου γνωμοδότησης. Ε, γύρεται λοιπόν το εξής ερώτημα. Η αναπτυξιακή διάσταση έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη σε αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία μεταξύ τεσσάρων χωρών αποτελεί φρένο για την περιφερειακή ολοκλήρωση, ναι ή όχι. Δεν έχω γνώμη, θα ήθελα την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, η ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σε αυτό το θέμα έχουμε ένα πρόβλημα που προκύπτει ξανά και ξανά. Τα άλλα κείμενα όπου περιλαμβάνονται ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, π.χ. η Σύμβαση του Κοτονού, αρκούν επαρκούν για να εξαναγκάσουμε μια χώρα με την οποία έχουμε συμφωνία ή συνάπτουμε συμφωνία αρκούν για να εξαναγκάσουμε αυτή τη χώρα να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν το γνωρίζω. Ναι ή όχι δηλαδή. Εάν όντως αρκεί, από τη στιγμή που έχει εγγραφεί σε προηγούμενο κείμενο και άρα είναι υποχρέωση που είναι ήδη σε ισχύ, πρέπει κάθε φορά να επανερχόμεθα πάνω σε μια τέτοια διάταξη και ρήτρα περί ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ή είναι πλεονασμός αυτό, ή είναι λίγο ε, κοροϊδία θα έλεγα, γιατί είτε ε, γίνεται σεβαστή η ρήτρα αυτή ήδη από τα προηγούμενα έγγραφα που ισχύουν, είτε δεν γίνεται ούτως ή άλλως. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι προβλέπει η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού. Και Έχουμε όντως μπροστά μας ένα πραγματικό πρόβλημα και το κακό έγινε πριν από καμιά δεκαριά χρόνια όταν ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση δίδοντας προτεραιότητα στο εμπόριο ο Επίτροπος Μάντελσον τότε είχε ξεκινήσει να διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ ο Επίτροπος για την Ανάπτυξη ξεκάθαρα είχε πει ότι οι συμφωνίες οικονομικής περιφερειακής εταιρικής σχέσης να είναι αναπτυξιακές συμφωνίες. Δηλαδή ο Επίτροπος για τα αναπτυξιακά θέματα έπρεπε να είχε πάρει αυτό το φάκελο και επειδή δεν του ανατέθηκε η αρμοδιότητα είχε πολύ λιγότερες δυνατότητες παρέμβασης τελικά. Έχετε λοιπόν την εντύπωση ότι μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει καλύτερα εδώ και δέκα χρόνια εάν εξ αρχής είχαν, ήταν σε ισότιμη βάση οι δύο επίτροποι. Αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τελευταία ερώτηση. Ο εισηγητής μιλά για απώλειες στον προϋπολογισμό που δεν αντισταθμίζονται. Μπορεί η Επιτροπή να μας πει ποιες είναι οι δυνατότητες ίσπραξης ε, των ε, δημοσιονομικών απολειών και αν ε, έχει ληφθεί υπόψη μια τέτοια δυνατότητα. Γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, μπορούμε πράγματι να πάμε πολύ μακριά ως προς την αντιστάθμιση, για τις απώλειες που έχουμε υποστεί. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαρτίνεθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ γνωρίζω το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο κύριος Γκέρενς βεβαίως και όλοι εμείς που το γνωρίζουμε ξέρουμε πώς ξεκίνησε στραβά το θέμα αυτό, διότι ο Επίτροπος που ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση την ξεκίνησε σε εσφαλμένη βάση, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο, για να μην πω και τίποτα χειρότερο. Η κυρία Άστον τους λίγους αυτούς μήνες με μετά την ε, ανάληψη των καθηκόντων της πράγματι σημείωσε πρόοδο. Πολύ σημαντική. Άκουσε όλους τους ε, συνομιλητές. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Όλα αυτά είναι αποδεκτά και συμφωνώ με όλα αυτά. Με το εξή δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ποιο. Άπαξ και υπογράφεται μία συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία, με τους Αφρικανούς συνομιλητές μας. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε ε, κατά κράτος πατερναλιστές και να πούμε ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Αφρικανών γιατί αυτοί δεν ξέρουν πώς να υπερασπιστούν τα δικά τους. Εάν οι συνομιλητές μας από την Αφρική υπογράφουν την συμφωνία τότε για λόγους σεβασμού απέναντί τους δεν μπορούμε να τους ε, μεταχειριζόμαστε ως κακομύριδες και ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα από αυτούς με μια πατερναλιστική έτσι, άποψη και θεώρηση της κατάστασης. Εγώ ήμουν μάρτυρα της υπογραφής συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Καραϊβικής Φτάσαμε στην κοινοβουλευτική συνάντηση ε, τρέφοντας αυτά τα αισθήματα για αυτούς τους κακομύριδες που τους είχαμε στρίψει τον αγώνα και τους είχαμε εξαναγκάσει να προσέλθουν στη συμφωνία και ούτω καθεξής. Και είδαμε ανθρώπους πολύ καλά ενημερωμένους που ήξεραν πολύ καλά τι ήθελαν και μας είπαν λοιπόν οι συνάδελφοι από την Καραϊβική ότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε, μελετήσαμε σε βάθος τη συμφωνία, βεβαίως έχει αρνητικά για μας όπως κάθε συμφωνία έχει και αρνητικά, αλλά υπάρχουν θέματα που μας ενδιαφέρουν και θα δούμε κατά πόσο είναι θετική ε, και θα την υπογράψουμε και βοηθά τα συμφέροντά μας και τα εξυπηρετεί. Ενώ συνέχιζαν οι διάφοροι από μη κυβερνητικέ οργανώσει και λοιποί να λένε ότι εμεί εξαναγκάζαμε ε, την ε, φτωχολογιά τη Καραϊβική. Ενώ δεν ίσχυε καθόλου κάτι τέτοιο και δεν το παραδεχόντουσαν ούτε οι ίδιοι, δηλαδή αναλάμβαναν πλήρω τι ευθύνε του. Το ίδιο ισχύει και για την Αφρική. Αφού υπογράφουν, δεν μπορούμε συνεχώ να λέμε ε, ότι αυτοί δεν ξέρουν τι λένε και δεν ξέρουν και τι υπογράφουν επειδή είναι από την Αφρική. Υπάρχουν κάποια όρια και πρέπει να τα χαράξουμε και δεν πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μία συμφωνία είναι αρνητική για εμάς. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μία συμφωνία την οποία θεωρούν οι Αφρικανοί θετική για τους ίδιους, να πούμε εμείς ότι όχι δεν είναι θετική για σας γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα από εσά. Αυτή είναι μια πατερναλιστική συμπεριφορά για να μην την ονομάσω και απεικιοκρατική και για να μην την ονομάσω και υπεραιαλιστική μπορώ να πω αν κάτι μου ταιριάζει, αν συμφωνώ με κάτι, αλλά δεν μπορώ να πω αν ταιριάζει στον άλλον ή ότι όχι δεν ταιριάζει στον άλλον ενώ του άλλου του αρέσει πράγματι. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εκπροσωπεί η κυρία Γιάννα Πόπελκόβε από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Χαίρομαι που μπορούμε να εκφράσουμε και εμεί τις απόψεις μας εδώ, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει τα σχόλιά σας πάρα πολύ στα σοβαρά. Η συμφωνία, όπως ξέρετε, είναι η πρώτη που εφαρμόζεται στην Αφρική. Γι' αυτό η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει με αυτή την ευκαιρία να αναφέρω κάποια θέματα που περιλαμβάνονται και στη γνωμοδότηση και θέλω να διασκεδάσω κάποιες ανησυχίες σας επίσης. Είναι κρίμα που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι από τις τέσσερις χώρες που υπέγραψαν, γιατί είμαι βεβαία ότι θα επαναλάμβαναν την ευνοϊκή θέση που εξέφρασαν στην πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή ΙΤΠΑ, αλλά και στη δική μας συνάντηση την εσωτερική που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Και οι τέσσερις χώρες σαφώς ε, τάχθηκαν υπέρ συμφωνιών σε μακροπρόθεσμη σταθερή προβλέψιμη βάση και ο εκπρόσωπος της Μαδαγασκάρης επανέλαβε τη θέση του και τη θέση της χώρας του ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να πάνε πέρα από το, τις συμφωνίες ΕΜΠΑ, οτιδήποτε εκτός από όπλα και θέλουν να στηρίξουν τη σχέση τους ε, πάνω σε κάτι πιο διατηρήσιμο και προβλέψιμο. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μαρτίνες γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφισβητούμε ε, υγιείς και καλές αποφάσεις ε, κυρίαρχων χωρών και νομίζω ότι καλύτερα θα κάνουμε να ψάξουμε τρόπους για να στηρίξουμε τους εταίρους μας στη διαδικασία υλοποίησης. Αργότερα θα δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου που είναι υπεύθυνη για την αναπτυξιακή συνεργασία που θα εξηγήσει λεπτομερέστερα τι μπορούμε να κάνουμε για τις χώρες αυτές. Ε, να πω ορισμένα πράγματα για τις ε, διαπραγματεύσεις είπα. Η Ανατολική μας Σημερινή Αφρική είναι δύσκολη περιοχή, ετερογενής και αυτό σημαίνει προκλήσεις για τις διαπραγματεύσεις. Όμως εμείς τις ε, ετερογένειες και τις διαφορές τις λαμβάνουμε πλήρως υπόψη όταν διαπραγματευόμαστε με αυτές τις χώρες και προσπαθούμε να τις λάβουμε υπόψη και να είμαστε και έλικτοι και να λάβουμε υπόψη μας και να καλύψουμε τις διαφορές να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ένα παράδειγμα ευελιξίας είναι η ασύμετρη προσέγγιση στο επίπεδο της απελευθέρωσης. Όπως βλέπετε, οι Σεϊχέλες και ο Μαυρίκιος προχώρησαν πολύ περισσότερο από το 90% στην απελευθέρωση. Δική τους απόφαση ήταν, ενώ η Ζιμπάμπου και η Μαδαγασκάρη, που είναι λιγότερες, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αποφάσισαν να απελευθερώσουν το 80%. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε ε, και να λάβουν υπόψη μας τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Ένα στοιχείο όμως ε, στο οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς είναι η καλή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και ο σεβασμός σε αυτά. Και υπάρχει σαφή σχέση με αυτά και με τη συμφωνία, γιατί συνδέονται και με τη συμφωνία του Κοτονού στο άρθρο 65. Οπότε υπάρχει η ρήτρα μη υποχρέωσης, μη εκτέλεσης, ε, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα για να πιέσουμε τις χώρες αν δεν συμφωνούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια λέξη για την βιώσιμη ανάπτυξη. Διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία πλήρη και συνεκτική με τις χώρες της περιοχής και συμφωνήσαμε με τις χώρες αυτές να καλύψουμε και την εργασία και το περιβάλλον. Αυτό θα είναι μέρος του συνολικού πακέτου όταν συμφωνηθεί. Και οι δύο πλευρές έχουν λάβει αυτή την υποχρέωση. Κύριε Κιόρενς, Κομισιό, με συγχωρείτε, σας εγκαλώ ως προς δεξής. Συμφωνώ με τον Μαρτίνες ως προς την αποδοχή από τους Αφρικανούς της συμφωνίας. Αυτές οι τέσσερις χώρες την απεδέχθησαν, εκεί δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Το πολιτικό μου ζήτημα δεν βρίσκεται εκεί. Το θέμα είναι γιατί οι άλλες χώρες δεν υπέγραψαν. Εξού και ο χαρακτήρα τη πρόθεση σε περιφερειακό επίπεδο. Η Κομισιόν θα μας πει γιατί οι άλλες χώρες δεν συνυπέραψαν την συμφωνία. Κομισιόν, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ένα, μισή λεπτό για την απάντησή σας, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Οι άλλες χώρες, εν συντομία, αποφάσισαν να αντιπραγματευτούν το πλήρες πακέτο. Το πλήρες τελικό πακέτο που αυτή τη στιγμή είναι υπό διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η βασική απάντησή μου. υπάρχουν μερικές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες οι οποίε διαπραγματεύονται καλύτερου όρου σε σχέση με το παρελθόν. Είναι κυρίαρχη η αποφασή του να παρέλθουν και να διαπραγματευτούν, επαναλαμβάνω, επί τη βάση ενό μεγαλύτερου συνολικότερου τελικού πακέτου. Παρακαλώ. Για να καταλήξουμε κάπου, Από ό,τι βλέπω υπέγραψαν μόνο τέσσερις χώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν τις κατηγορίες περί εμπεριαλισμού. Το βασικό εδώ είναι το εξή. Έχουμε 16 χώρες στην αρχή. Τέσσερις μόνο συνυπογράφουν. Πώς είναι δυνατόν οι άλλες να μην ακολουθούν και να προσπαθούν να διαπραγματευτούν ένα ευρύτερο πακέτο. Δεν μπορώ να καταλάβω τα κίνητρά τους. Τώρα, άκουσα ότι πρόκειται περί τροπολογιών. Δεν ξέρω τι, τι μπορεί να κάνουμε με τις τροπολογίες. Το θέμα είναι ναι ή όχι. Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Η Γιούριτ είπε να μην συνενέσουμε. Υπάρχουν φυσικά και άλλα επιχειρήματα, υπάρχει και κατά. Να τα ακούσουμε για να πάρουμε και μία απόφαση τελικά. Η Γιούριθ πάντως, το καταγράφω αυτό, λέει όχι. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Κατάθεση τροπολογιών ως τις 14 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στις 6 Δεκεμβρίου. Και τώρα, Σημείο 14. Επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα δικαιώματα του ανθρώπου. Ο κ. Κέιτ Τέιλορ είναι ο εισήγητης. Κίθ, έχεις τον λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομος λόγω της καθυστέρησης για την οποία βεβαίως είμαι υπεύθυνη. I'm sorry, Chair. Without Συγγνώμη. Ανεφετέρας, σας ευχαριστώ και θα είμαι και όσο πιο σύντομος μπορώ. Αλλά είναι σημαντικό το θέμα γιατί η χρηματοπιστωτική κρίση έχει γίνει διεθνής και ε, έχει διαφορετική ένταση ανάλογα με το αν ε, έχουμε και επισητιστική κρίση κλπ. Δύσκολα κάνουμε γενικεύσεις λοιπόν. Στην Ανατολική Ασία ε, πέρασε στο εμπόριο και τις αγορές εργασίας η κρίση. Στην υποσαχάρια περιοχή, στο Ανατολικό Ιρωνικό ε, τα προβλήματα ήταν στις εξαγωγές βασικών αγαθών, στις μειώσεις δασμών. Στη Λατινική Αμερική δυστυχώς φαίνεται ότι είχαν και τα δύο. Τα πάθαν και τα δύο. Αλλά ε, υπάρχουν ε, ε, προβλήματα ρευστότητα για τις κυβερνήσεις που προσπαθούν να, του, να, τις, να στηρίξουν όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι σαφές ότι η κρίση είχε και κοινωνικό αντίκτυπο και οικονομικό. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας υπολογίζει ότι οι καταγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 20 εκατομμύρια και περισσότερο μέχρι το τέλος του 2009 και υπάρχουν και μερικά ακόμη εκατομμύρια άνεργων που ε, αναγκάστηκαν να πάρουν επισφαλείς θέσεις εργασίας και αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στις επίσημες στατιστικές ανεργίας. Ο αναπτυξιακός στόχος της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους τώρα υπονομεύεται. Αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη διαρθρωτική και δομική πρόοδος, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη κοινωνική προστασία και να ανταποκριθούμε στην καθολική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίως λόγω της κρίσης, η Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Εθνή υπολογίζουν ότι μεταξύ 55 και 103 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Και η μείωση της ε, φτώχειας στην υποσαχάρια ε, Αφρική επιβραδύνεται τώρα. Και μεταξύ 30 και 50 χιλιάδες περισσότερα παιδιά πέθαναν σε αυτή την περιοχή το 2009 ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση εφιστώ την προσοχή στις δυσκολίες στην πρακτική επιβολή και παροχή οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων παρά ότι το γεγονός ότι οι διεθνείς κοινότητες αναγνωρίζουν το αδιέρετο και την ίση σημασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Διεθνή Συμφωνία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, οικονομικά και κοινωνικά που επιτρέπουν καταγγελίες ε, αν υπάρξουν παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων. Νομίζω ότι η απουσία πολιτικής λογοδοσίας ε, για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, για τα πολιτισμικά, επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική κρίση. Αυτό που άρχισε ως ε, χρηματοπιστωτική κρίση, γρήγορα ε, έγινε κρίση των παγκοσμίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταρχήν βλέπουμε ότι τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα παραβιάζονται γιατί και υπάρχει ένας φαύλος ε, κύκλος ε, ο οποίος ε, τάσεται κατά των ξένων και δημιουργεί ξενοφοβία και έτσι οι ξένοι δεν μπορούν να βρουν καλές, καλή δουλειά. Επίσης μειώθηκαν τα εμβάσματα στον κόσμο, τα μειωμένα εμβάσματα και τα μειωμένα εισοδήματα των οικοκαιριών απειλούν την ε, ήδη εύθραυστη επιβίωση αυτών των πολλών οικογενειών. Επίσης, τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα υπονομεύονται και το δικαίωμα στην τροφή, στα τρόφιμα, που αυξάνει την φτώχεια και κάνει τους ανθρώπους να μειώσουν την ποιότητα και ποσότητα της διατροφής. Τα δικαιώματα στην υγεία ε, υπονομεύονται. 400.000 ε, περισσότερα βρέφη θα πεθάνουν κάθε χρόνο ως συνέπεια της κρίσης αυτής, σύμφωνα με την UNESCO. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην παιδεία, ιδιαίτερα την εκπαίδευση των γυναικών, απειλείται γιατί οι οικογένειες δεν, μπορεί, δεν έχουν την πολυτέλεια να στείλουν τα κορίτσια τους στο σχολείο και τις βάζουν να κάνουν οικιακά ή χαμηλόμιστες ε, ε, θέσεις εργασίας. Ε, επίσης, οι μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας ε, κάμπτονται και αυτό αυξάνει τη φτώχεια. Επίσης, η επίδραση στο κοινωνικό φύλλο επηρεάζεται ε, και αυτό, γιατί οι γυναίκες πολλές φορές ε, είναι σαν εφεδρικό στρατός ε, στην κρίση και ε, όλα τα προβλήματα αυξάνονται. Είναι πιο πιθανό επίσης να αντιμετωπίσουν αυξημένη οικογενειακή βία, σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπορία αυξάνεται η απλήρωτη εργασία για τις γυναίκες και αυτό έχει πολλές επιπτώσεις στα δικαιώματά τους. Είναι ζωτική σημασία να θυμόμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν παρεκκλήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα και σε περιόδους κρίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα καθολικά εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Οι κυβερνήσεις έχουν άμεση ευθύνη να διασφαλίζουν ε, ελάχιστα ουσιώδη επίπεδα κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων. Θα μπορούσα να μιλήσω κι άλλο, κυρία Πρόεδρε, αλλά μου φαίνεται ότι ε, πιέζει ο χρόνος. Θα πρέπει να δούμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε δημοσιονομικά μέτρα, θέματα διαφάνειας, κυρίως στην Αφρική, την ανάγκη για διαφάνεια. Θα πρέπει να ε, γίνουν ε, δημοσιονομική έλεγχη και φορολογική έλεγχοι στις χώρες αυτές για να ξέρουμε πολύ καλά πού πάνε και από πού έρχονται τα χρήματα. Ε, αν δούμε την νεοφιλελεύθερη δομή του εμπορίου, έτσι όπως αναπτύχθηκε, βλέπουμε ότι αυτό ακριβώς είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα στις συζητήσεις ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της, η μεγέθυνση από μόνη της, δεν εγγυάται ωφέλη για τους φτωχούς. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Ήμουν στην Επιτροπή Ίντα τα προηγούμενα δύο χρόνια και μπορώ να σας πω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι σε δεύτερη θέση. Πρώτο είναι το εμπόριο. Θα πρέπει να έχουμε μια συνοχή στην ε, αναπτυξιακή πολιτική. Περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις είναι υποψήφιοι μιλητές. Παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας. Λόγω του προκεχωρημένου της ώρας. Δύο λεπτά νομίζω είναι υπεραρκετά. Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος του σκιώδου συζητητή του κυρίου Κάσμαν. Καταρχάς ευχαριστούμε τον κύριο Τέιλορ για την ε, γνώμη που εξέφρασε, για την γνωμοδότηση, για την αναφορά στην καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως εργασιακών δικαιωμάτων. Η κρίση αυτή τη στιγμή ε, φέρει μεγάλο πλήγμα σε τέτοιου είδους οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία όμως τίθενται στο περιθώριο, πίσω από τις ε, από τα στοιχεία του ΑΕΠ πίσω από την κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηρίων κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι ε, υποφέρουν. Και εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες έτσι ώστε το κείμενο αυτό να είναι πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς και να μιλήσουμε και για τα εργασιακά ε, προβλήματα των μειονοτήτων. Θα μιλήσουμε για την διασφάλιση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δυνατότητα να χαλιβδοθούν όλα αυτά τα εργασιακά και εκτιμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρενς. Ε, Συμφωνώ με την ανάλυση του κύριου Τέιλορ. Παρ' όλα αυτά, να έχει υπόψη του το εξή. Πιστεύω ότι η οικονομική κρίση, η χρηματοοικονομική και η οικονομική κρίση δεν φταίει για την επιδείνωση της κατάστασης των δικαιωμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το πρόβλημα χρονολογείται από παλαιότερα. Σύμφωνα με την Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεω, Τα πήγε καλά η Αφρική στην κρίση. Συνέχισε να αναπτύσσεται με ρυθμούς περίπου 5%. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε για τα προβλήματα που έθιξε ο κ. Τέιλορ. Λοιπόν, ε, όπω είπε και ο Μπουρλάος, έχουμε στα χέρια μας ένα μαχαίρι το οποίο έχει λάμα αλλά δεν έχει λαβή. Στο G20, κοιτάξτε, δεν πάμε καλά. Ε, τα αποτελέσματα παρά τις προσπάθειες είναι σχεδόν μηδενικά. Πιστεύω καταρχήν ότι πρέπει να κωδικοποιήσουμε τα δικαιώματα, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το μέσο είναι η πολιτική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς της Κομισιόν. Πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε οι σχέσεις μας να είναι φιλόδοξες, απαιτητικές, πρέπει να είναι οι καλύτερε Έτσι μόνο θα προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε έξυπνου τρόπου συνεργασία. Και αυτό σίγουρα δεν μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να σωματώσουμε στα διάφορα κείμενα, μέτρα, ε, δεσμευτικά υπέρ των δικαιωμάτων. Πρόκειται, εν πάση περιπτώσει, για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, το βλέπουμε και προκειμένου, αλλά και στις προηγούμενε τρει με τέσσερι εκθέσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριο Γκούστευσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να πω αρχικά ότι είναι εξαιρετική πρόταση με πολύ καλά συστατικά. Με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με ε, ηθικό τρόπο προσεγγίσατε τα θέματα. Το μόνο που θα προσέθετα είναι ότι υπάρχει έλλειψη της προοπτικής της ισότητας, αλλά στην προφορική σας παρουσίαση, πολύ σωστά, είπατε, μιλήσατε για τη σχέση αυτή. Αν υπάρχουν απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, συνήθως τα γυναικεία ανθρώπινα δικαιώματα θίγονται πιο πολύ από εκείνα των ανδρών. Αυτό να το αναδείξουμε, να το καταδείξουμε και να το συμπεριλάβουμε στην ανάλυση μας. Και χαίρομαι που τα είπατε και το, μιλήσατε και για τα γυναικεία ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. Το μόνο που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε είναι να βάλουμε αυτήν την ε, παράμετρο στην πρόταση και να ακολουθήσουμε το πνεύμα της ε, παρουσίασής σας. Και να το βάλουμε και να είναι και γραπτός. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δεν ξέρω ποιος την εκπροσωπεί όμως. Δύο λεπτά και πάλι παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Πρόεδρε, είμαι ο Μάικλ Σουάν στην, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχω να κάνω κάποια ιδιαίτερη δήλωση. Μόλις ε, ήρθα από την Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου έγινε πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεσης και επιβεβαιώνω αυτό που είπα και εκεί, ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα προφανώς και επειδή λάβαμε τώρα μόλις την έκθεση τις ε, τελευταίες ημέρες, θα, τις, θα τη μελετήσουμε για να παρουσιάσουμε μία έγκυρη ε, άποψη. Το μόνο που είπα στην ε, υποεπιτροπή και που θα έπρεπε, θα ήταν ενδιαφέρον να αναφέρεται και στην έκθεση και φυσικά και στον προβληματισμό αυτής της Επιτροπής είναι η ανάγκη να δούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την λήξη του ορίζοντα του 2015 για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Γιατί εκεί θα χρειαστεί πολύ σημαντική μελέτη από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη-μέλη. Είμαστε στα, στην πρώιμη φάση αυτής της διαδικασίας, αλλά ξέρουμε και από προηγούμενα τέτοια εγχειρήματα ότι ο χρόνος θα μας πιέσει πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Κύριε Τέιλορ, να κλείσουμε. Έχετε το λόγο. Στα γρήγορα, ευχαριστώ πολύ για τα θετικά σας σχόλια. Συμφωνώ απόλυτα ότι ένα πράγμα είναι να κατανοούμε το πρόβλημα που αφορά την εξασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλο πράγμα είναι να βρούμε λύση για το πρόβλημα. Γι' αυτό χαιρετίζω ιδιαίτερα την ιδέα μιας εταιρική σχέσης εδώ. Μίλησα για την ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, μια Τετάρτη είναι. Κάποια πράγματα που αναφέρατε θα ε, κατατεθούν ως ε, τροπολογίες. Στην συνάντηση της ε, Ρώμης μιλήσαμε για την ασφάλεια των τροφίμων και μιλήσαμε και για τον ρόλο των γυναικών ε, ε, που τονώνουν τις τοπικές κοινότητες. Και ένας υπουργός από την Αιθιοπία είπε μάλιστα «Αλήθεια, πρέπει να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και τις κοπέλες, γιατί αυτό σημαίνει ότι ενδυναμώνουμε την κοινωνία και το μέλλον μας. Μην το ξεχνάμε αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες δεν θα είναι σε μειονεκτική θέση, γιατί παίζουν ρόλο βασικό στη κοινωνία. Και περιμένω τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υποβολή. Τροπο... Ε, ε, Αυτό... 8 Δεκεμβρίου. Ψηφίζουμε. Ε, περάμε μάλλον στις ψηφορίες. Να κάνουμε μια δοκιμή με τις κάρτες σας. Έναρξη ψηφορίας. Δοκιμάστε παρακαλώ τις κάρτες σας. Ε, λείπουν 7 ακόμη. Voilà, cartes Λείπουν ακόμη πέντε. Τρεις ακόμη. Δύο. Μία. Il manque trois. Μας λείπουν ακόμη τρεις ε, κάρτες. Τρεις κάρτες δεν φαίνονται εδώ. Ωραία. Ε, άλλη μία λείπει. Πέρας ψηφοφορίας. Συνεπώς, ειδική έκθεση αποτελεσματικότητα αναπτυξιακής βοήθειας έκθεση του κ. Σαλόμ. Τροπολογία 1. Να κάνουμε να ψηφίσουμε block ε, τις 1, 2 και 3 τροπολογίες. 1, 2 και 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Επί της ε, έκθεσης έλεξης ψηφοφορίας πέρα. Πέρασε. Εγκρίνεται ομοφόνος. έκθεση του κυρίου Νίκ. τροπολογία 1, υπέρ. Ψήσουμε ομαδικά τις, τις τρεις πρώτες, 1, 2 και 3, όχι. Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός την έκθεση στο σύνολό της έναρξη υπέρ πέρας. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται ομοφόνος. 24 ψήφοι. Της κυρία Στρίφλερ, στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για το της Αφρικής. Ψηφίζουμε on block. Όχι. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω όχι. Επιβεβαιώνουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Υπέρ. Έναρξη. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται 14 υπέρ 10 κατά. Τροπολογία 2 υπέρ. Τι υπόλοιπε μαζί. Οι 2, 3 και 4 λοιπόν. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε λοιπόν επί ε, έκθεσης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23 υπέρ μία κατά. Ψηφίσουμε τώρα για την... Ε, α, Μία ε, Μίας πέντε λέει κάποιος όχι, δεν μπορούμε. Τροπολογία 1 στο επόμενο. Ερώτηση. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Α, να ψηφίσουμε μαζί τις 2, 3, 4 και 5. Ωραία. Μάλλον 2, 3 και 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία η τρία είναι σε τρία τμήματα. Για το πρώτο. Η πέντε με συγχωρείτε είναι. είναι σε τρία τμήματα. Δεύτερο τμήμα της πέντε, Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχές, Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα του, της πέντε, Υπέρ. Κατά. αποχές, Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την προφορική ερώτηση, την τροποποιημένη έναρξη ψηφορίας. Μας λείπει μία ψήφος. Πέρας. Ψηφορίας. Εγκρίνεται. Δεν έχουμε κάτι στα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίασή μας. 5η 6 Δεκεμβρίου, 9 με 12.30 και την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου από τις 3 ως τις 6.30 και την Τρίτη 18 από τις 9 έως τις 12.30 και από τις 3 έως τις 6.30. Μετά από αυτό, μια αντιπροσωπεία θα φύγει το Πελαμόντε. Συνεχίζουμε και κλεισμένα των θυρών και ο Σπέρμεν θα μας ενημερώσει για την τελευταία διαπραγμάτευση για τον μηχανισμό αναπτυξιακής εργασίας. DCI. Παρακαλώ λοιπόν, ε, ώστε την Εμέλη να βγουν από την αίθουσα.